Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζουμε. Συνεδρίες Επιτροπής μας, τα γνωστά σημεία. Πρώτο σημείο, έγκριση μερίσης διάταξης που έχει κυκλοφορήσει. Δεν διαφωνεί κανείς. Εγκρίνεται η μερίσια διάταξη και προχωρούμε σημείο 2, ανακοινώσει του Πρόεδρου. Καμία για εξαίρεση. Και πάμε αμέσω στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Τα έχετε τα πρακτικά. Ε, και μάλλον συμφωνείτε γιατί έχουν συζητηθεί τα πρακτικά προηγουμένω. Και αν δεν διαφωνήσει κανείς και καθώς δεν διαφωνεί προχωρούμε αμέσως στο σημείο υπεριθμών 4. Έχουμε εδώ την ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010. Θα ακολουθήσει παρουσίαση από τον αρμόδιο τον οργανισμό των θεμελιδών δικαιωμάτων, τον κύριο Μόρτεν Τζέρουμ. Τον καλωσορίζουμε. Σήμερα το πρωί, συνεδρίασή σήμερα, για να μας παρουσιάσει την ετήσια έκθεση για το 2010 agency που μόλις εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του κανονισμού του Συμβουλίου ε, πρέπει να παρουσιαστεί στην Επιτροπή μας. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Θεμελιώδη δικαιώματα, προκλήσεις και επιτεύγματα». Αναλύει την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στους τομείς που καλύπτει ο οργανισμός στο πολιετές του πρόγραμμα. Η έκθεση συνοδεύεται και από μία σύνοψη με τίτλο «Κομικά σημεία για τα θεμελιώδη δικαιώματα και εξελίξεις το 2010». Υπάρχει στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα πολωνικά και στα ουγγρικά. Θα ακούσουμε λοιπόν το Διευθυντή, τον κύριο Τσέρουμ και στη συνέχεια θα ε, ακολουθήσει συζήτηση. Έχετε το λόγο κύριε Διευθυντά. Μετά θα ακούσουμε και την κυρία Μπραντς Κέρις. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται ενώπιον της Επιτροπής μας. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Α, πρώτα η κυρία Κέρις τότε. Η κυρία Μπραντς Κέρις πρώτη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι προνόμιο και τιμή για μένα ευκαιρία που έχουμε να έρθουμε ενώπιον σας να σας παρουσιάσουμε την ετήσια έκθεση του οργανισμού μας για τις προκλήσεις και τα επιγεύματα του 2010. Φαντάζομαι έχετε ήδη την έκθεση στα χέρια σας. Είναι περίπου 200 σελίδες φέτος. Ε, είναι πολύ βαριά η έκθεση αυτή, με πολλές έννοιες και ελπίζω να ε, έχετε την ευκαιρία να τη χρησιμοποιείτε στις εργασίες σας. Η έκθεση αυτή είναι τόσο μακροσκελής, όχι για να ζυγίζει, αλλά ε, το βάρος της είναι ειδικό βάρος και σημαντικό για να βοηθήσει ε, στην περαιτέρω εργασία μας και μάλιστα συνεργασία μας για την πρόθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι μια επισκόπηση των προκλήσεων, των πρακτικών, των προβλημάτων και θα συζητήσουμε θέματα που έρχονται από το άσυλο, την προστασία των δεδομένων, δικαιώματα των παιδιών, δικαιώματα μειονοτήτων. Από τότε που καταθέσαμε την ετήσια έκθεση πέρυσι, οι σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Οργανισμού συνεχίζουν να διευρύνονται και να εμβαθύνονται και θα ήθελα να σας δώσω και μερικά παραδείγματα σχετικά. Πρώτον, κατόπιν αιτήματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόσφατα γνωμοδοτήσαμε δύο φορέ ε, για θέματα ποινικού δικαίου. Η πρώτη γνωμοδότηση ήταν το Φεβρουάριο για το την Ευρωπαϊκή Εντολή Ερεύνης ε, και το δεύτερο ήταν για το PNR. Και ε, ε, απεστάλλει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τα δύο έχουν να κάνουν με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την ιδιωτική ζωή, καθώς αυξάνεται η διακρατική συνεργασία στο ποινικό δίκαιο. Ένα δεύτερο παράδειγμα της συνεργασίας μας του Φεβρουαρίου είναι ότι με μεγάλη χαρά ε, παρουσιάσαμε με μια ε, εγκυκλοπαίδεια Charterpedia ε, σχετικά με το χάρτη των θεμελιδών δικαιωμάτων και βασίζεται και πάλι στη δική σας δουλειά και την προσφέρουμε κατόπιν δικού συστήματος. Επίσης, Άλλη ένδειξη των αναπτυσσόμενων σχέσεων μας είναι η συνειδητοποίηση ε, της εργασίας του κάθε οργάνου και οργανισμού. Και αυτό ε, είναι σημαντικό. 11 ε, φορές αναφερόμαστε σε έγγραφά μας σε δικά σας ψηφίσματα. Και αυτό όλο και πιο σημαντικό. Είναι λοιπόν μεγάλη η προσοχή που δίνεται σε αυτά τα θέματα και πάγια και διαρκή. και αυτό σημαίνει ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό να εκδίδεται αυτή η ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, είναι πολλές οι λειτουργίες και οι σκοποί που εξυπηρετεί. Ο πρώτο είναι ότι μπορεί να είναι σημαντικό σημείο αναφορά. Για παράδειγμα, όταν συζητάτε την οδηγία για τα θύματα, ε, θα δείτε ένα κεφάλαιο για την αποζημίωση των θυμάτων ε, αξιόπινων ε, πράξεων και περιλαμβάνει εθνικές, διεθνείς, ευρωπαϊκές εξελίξεις, παραδείγματα. Ελπίζω να έχετε την ευκαιρία να μελετήσετε την έκθεση αυτή. δεύτερη αποστολή, ας πούμε, η μία από τις άλλες αποστολές της είναι έρευνα που μπορεί να υποστηρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που, όταν κάνουν τα, τις δικές τους εκθέσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ξέρω ότι ε, και οι εκθέσεις αυτές ε, είναι συμπληρωματικές και προσθέτουν. Οι εκθέσεις του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζουν ε, την πολιτική και δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές, ενώ εμείς έχουμε ως ρόλο να υποστηρίζουμε με ένα χάρτη ε, και τα δύο αυτά θεσμικά όργανα για να είναι ένας μπούσουλας, ας πούμε, για την καθημερινή του δουλειά. Εξετάζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κράτη-μέλη, βασιζόμαστε σε στοιχεία που συλλέγουν τα κράτη-μέλη και στέλνουν ε, αρμοδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση ε, τις εξελίξεις και τις διεθνείς. Τελειώνω την εισαγωγή μου λέγοντας ότι παρόλο που η εντολή μας είναι ευρεία, εμεί περιοριζόμαστε σε θέματα ε, που ορίζει το πολιετές μας πλαίσιο λειτουργίας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Το Κοινοβούλιο θα έχει την ευκαιρία βεβαίω στο μέλλον και ελπίζω σε ένα προσεχές μέλλον να διευρύνει το πολιετές πλαίσιο. Ε, θα έχει την ευκαιρία να το εξετάσει, ελπίζω, και θα συμπεριλάβει και την επανεξέταση των μελλοντικών θεμάτων για την επόμενη περίοδο 2013-2018. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι αποστολή μας να ασχολούμαστε και με τα θεσμικά όργανα και με τα κράτη-μέλη και να τους παρέχουμε βοήθεια και πραγματογνωμοσύνη για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εάν δεν αναθεωρηθεί το πολιετές μας πλαίσιο ε, για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις συνθήκης Λισαβόνας, μπορεί να υπάρξουν κενά ε, και προβλήματα και περιορισμοί στην εργασία μας. Προσβλέπω ε, στο μέλλον σε μια γόνιμη συνεργασία για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, χωρίς να χάνουμε το τελικό μας στόχο να απολαμβάνουν θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι όσοι διαμένουν σε αυτή. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον Διευθυντή του Οργανισμού, τον κύριο Μόρτον Κιάνουμ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you, Σας ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τον Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τον κύριο Κέρουμ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερος ε, που σας παρουσιάζω τα επιτεύγματα, τα φετινά επιτεύγματα του οργανισμού, όπως ε, αποκρισταλώνονται στην ετήσια μας έκθεση, που ελπίζω να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς και στο δικό σας έργο για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η ετήσια έκθεση ε, παρέχει στοιχεία και αναλύσεις για την κατάσταση θεμελιωδών δικαιωμάτων και στις 27 χώρες μέλη. Επισημαίνει τις ε, θεμελιώδεις εξελίξεις και τις σημαντικότερες προκλήσεις και στη χάραξη πολιτικής, αλλά και επί το καθημερινά. Επίσης, χρησιμοποιεί υποδείγματα κάποιες ελπιδοφόρες πρακτικές που μπορεί να χρησιμεύσουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρεις βασικούς κλάδους θεμελιώδων δικαιωμάτων από την φετινή ετήσια έκθεση που είναι ιδιαίτερα σημαντικά από πολιτική άποψη. Καταρχήν θέματα μετανάστευσης και ασύλου Δεύτερον, κατάσταση των Ρωμά. Και τρίτον, η αναπηρία στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτο σημείο, μετανάστευση και άσυλο. Η ετήσια έκθεση επισημαίνει τη μεταναστευτική πίεση που ασκείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που έχουν εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που οδήγησε σε μεγάλες δυσκολίες ό,τι αφορά την εξασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υποδοχής και το δικαίωμά τους για άσυλο. Έρευνες που έγιναν από τον οργανισμό μας επιτόπου βρήκαμε συνθήκες σε σε στρατόπεδα υποδοχής με ελεηνές υγειονομικές συνθήκες, χωρίς ζεστό νερό και μάλιστα σε αντίξου χειμώνες. Επίσης ε, δεν είχαν δυνατότητα αυτοί που έχριζαν προστασίες πραγματικά να υποβάλουν αίτηση για άσυλο. Δηλαδή, με βάση τον κανονισμό του Δουβλίνου 2, άνθρωποι που πραγματικά έπρεπε να χαίρουν προστασία, ε, δεν μπόρεσαν να την ασκήσουν. Το σύστημα ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίσει αποφυγή της, ε, του επαναπατρισμού εφόσον το κράτος υποδοχής δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα στοιχ, τις στοιχειώδεις προδιαγραφές θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μάλιστα, η πίεση επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένε χώρε των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δείχνει την ανάγκη περισσότερων μέτρων αλληλεγγύη ω τμήμα ενό ευρύτερου συστήματο προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα θέματα αυτά και οι επιπτώσει του για τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στι ε, συζητήσει για τη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασύλου. Δεύτερον, ασχολούμαστε με την εφαρμογή θεμελιωδών δικαιωμάτων στους Ρωμά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ετήσια μας έκθεση προ... επισημαίνουμε την προσπάθεια καταπολέμησης της περιθωριοποίηση αυτής της κοινότητα στο Ρωμά. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τι εθνικέ πολιτικέ ε, Ένταξης, φαίνεται ότι ε, θα πρέπει να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση στοιχείων για το θέμα αυτό. Στην ετήσια μα έκθεση τονίζουμε τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της κοινότητας των Ρωμά και του υπόλοιπου πληθυσμού. Βλέπουμε για παράδειγμα τα ποσοστά απασχόλησης για τους Ρωμά κυμαίνονται μεταξύ 10 και 30% ε, ήταν κατά 10% χαμηλότερα τα ποσοστά απασχόλησης από τα ποσοστά απασχόλησης του υπόλοιπου πληθυσμού στις χώρες που πραγματοποίησαμε έρευνα και θα συνεχίσουμε τις έρευνες όχι μόνο για την απασχόληση, αλλά και για την υγεία, την παιδεία και θα βρείτε πολύ περισσότερα στοιχεία στην ετήσια μας έκθεση. Τώρα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένες από τις προτάσεις που υποβάλλει ο οργανισμός μας στην ετήσια έκθεση, προκειμένου να ξεπεραστούν οι προκλήσεις και για τους Ρωμά. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή της ε, κοινοτικής νομοθεσία για την αποφυγή της διακριτικής μεταχείρισης, Την πλήρη εφαρμογή αυτή τη νομοθεσίας της Ένωσης. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι τοπικοί μηχανισμοί, για παράδειγμα τα διάφορα, οι διάφοροι φορείς των Εθνικών Ινστιτούτων και τους υπόλοιπους φορείς που στόχο έχουν την προστασία των Ρώμα. Θα πρέπει να ενισχυθούν όλοι αυτοί οι φορείς. Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται με τις ε, εθνικές αρχές αλλά και τις κοινωτικές. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή συντονισμός μεταξύ των διαφόρων επιπέδων. Και τρίτον, θα πρέπει τα διαθέσιμα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φτάνουν πραγματικά σε τοπικό επίπεδο. Κάτι που θα διευκολυνθεί από μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων τοπικού, εθνικού και κοινοτικού. Τέλος, ε, έχουμε στο ζήτημα της αναπηρίας. Το ψήφισμά σας για τα θεμελιώδη δικαιώματα του περασμένου Δεκεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, χαίρεται για τη συμπερίληψη παραρτήματος στην ετήσια έκθεση του 2010 που κάνει μια επισκόπηση των ε, συνθηκών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεσμεύουν τα κράτη-μέλη. Και μάλιστα το παράρτημα αυτό μετατράπηκε σε αυτοτελές κεφάλαιο της ετήσιας μα έκθεση. Πέρυσι το Δεκέμβριο προσθέθηκε μια νέα διάσταση στις διεθνείς υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κύρωσε την ε, συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ε, προσώπων με αναπηρία. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ε, συμβαλόμενο μέρος σε μια διεθνή συνθήκη και πρέπει πια η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρήσει την αναπηρία ως θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων και όχι μόνο ως ζήτημα κοινωνικής πολιτικής. Βέβαια και το θέμα αυτό έχει άμεση σχέση με το έργο της δικής σας Επιτροπής. Και οι συνεχείς προσπάθειες του οργανισμού μας ε, εξασφαλίζουν την πολιτική συμμετοχή, τις ε, διάφορες ηθίκες ε, σε φορείς, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την παθητική και ενεργετική νομιμοποίηση των αναπήρων και ούτω καθεξής. Ελπίζω να ληφθεί υπόψη από σας το κεφάλαιο αυτό στο καθημερινό σας έργο και στην νομοθετική σας προσπάθεια. Ο οργανισμός μας θα συνεχίσει να συγκεντρώνει και να αναλύει τα διάφορα στοιχεία και στο μέτρο που προχωρά το έργο μας θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε καλύτερα και τις διάφορες τάσεις ε, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι δεν θα έχουμε απλά στιγμιότυπα κατακαιρματισμένα της κατάστασης, αλλά μία δυναμική εικόνα για ένα δεδομένο διάστημα. Και έτσι θα διαπιστώνουμε κατά πόσο οι νομοθεσίες και οι πολιτικές όντως λειτουργούν και βελτιώνουν την κατάσταση ή κατά πόσο θα πρέπει να τροποποιηθούν ή να ε, λάβουν μια νέα κατεύθυνση ανάλογα με τις εξελίξεις και με τις προκλήσεις που δημιουργούνται. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε για αυτή τη συνοπτική παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Οργανισμού Θεμελιώδων Δικαιωμάτων. Άρχεται η συζήτηση. Πρώτος ζήτησε το λόγο ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Διευθυντή ε, του οργανισμού καθώς ε, και την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σίγουρα θα μελετήσουμε διεξοδικά αυτή την ε, εκτενή έκθεση. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του εσύλου, της μετανάστευσης και της ένταξης και σε τρεις συγκεκριμένε πτυχές. Το ένα αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα. Αναφέρεται στην έκθεση του 95% το 75% των συλλήψεων γίνονται στα σύνορα της Ελλάδας. Αναφέρεται όμως ότι τα ελληνικά συστήματα για τη διαχείριση των αιτήσεων ασύλου ε, βρίσκονται στα σπάργανα ακόμη ε, και εκφράζεται δυσπιστία και τρίτων χωρών σε ό,τι αφορά την ε, μεταφορά ετούντων άσυλων. Σημείο 2 οδηγία για, την, για τον επαναπατρισμό. Ποια είναι η κατάσταση ό,τι αφορά την εφαρμογή, γιατί αναφέρεται ότι 8 κράτη-μέλη ακόμη δεν έχουν προσδιορίσει τους χρόνους διοικητικής κράτησης. Θα ήθελα ένα σχόλιο για το σημείο αυτό. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τη μονάδας Ράμπιτς, ό,τι αφορά τα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, υπήρχε αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του συστήματος ό,τι αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σας ευχαριστούμε κύριε Διασδεμέρη. Κυρία Στάνοκα. Yes, thank you, uh, well, uh, first... Ευχαριστώ. Μία γενική ερώτηση προς τον κύριο Κέρο. Βλέπουμε εδώ στη δομή της ετήσιας έκθεσης σε κίτρινο χρώμα κάποιες δραστηριότητες του Οργανισμού θεμελιών Δικαιωμάτων. Ίσως να κάνω λάθος, αλλά βλέπω ότι ουσιαστικά οι δραστηριότητες σας περιορίζονται στην εκπόνηση εκθέσεων και στην οργάνωση συναντήσεων και συνεδριάσεων. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. έχει και άλλε δραστηριότητε. ο οργανισμό Θεμελιώδων Δικαιωμάτων ή περιορίζεται σε εκθέσεις για την οργάνωση συνεδριάσεων. Δεύτερη παρατήρησε περισσότερο παρά ερώτηση. Το ίδιο ισχύει και για την περσινή σας άλλωστε ετήσια έκθεση. Και το βλέπουμε και στη φετινή. Ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν ε, ο οργανισμός σας δεν θεωρεί τους απάτριδες ή την ε, κατάσταση των απάτριδων ως ε, καταστρατήγηση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων ή ως μη διακριτική μεταχείριση. Είδε τη θεωρία ως περίπτωση της ε, παραβίασης της αρχής για μη διακριτική μεταχείριση. Γιατί... Ε, γιατί είναι μεγάλος ο πληθυσμός των απάτριδων, ειδικά στις βελτικές χώρες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ε, υπήκοοι κανένας κράτους και δεν ε, δικαιούνται να ψηφίσουν καν στις τοπικές, στις δημοτικές εκλογές, ούτε και στις ευρωεκλογές. Ακόμη και μιλούμε για υπηκόστριτων χωρών, καλό θα ήταν να γίνει στο αντίστοιχο κεφάλαιο της δημοκρατικής συμμετοχής μια ανάλυση. Είπατε ότι δεν έχετε δεδομένα για το πόσοι, πόσοι εξοκοινοτικοί συμμετέχουν, ε, διαμένουν και λαμβάνουν μέρος σε εκλογές. Πάντως, πολλά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνουν συστάσεις για την συμμετοχή των μονίμων κατοίκων στις εκλογές. Ίσως ε, καλό θα ήταν ο δικός σας οργανισμός να κάνει μια απογραφή της κατάστασης, να κάνει μια έρευνα για το βαθμό του προβλήματος σε διάφορα κράτη-μέλη. Ερωτώ λοιπόν, θα ήταν σε θέση ο οργανισμός να διεξαγάγει μια τέτοια έρευνα και να μην επικαλείται απλώς την έλλειψη χορηγής στοιχείων από τα κράτη-μέλη. Η κυρία Γκυγιόμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για αυτή την διεξοδική παρουσίαση που μας δείχνει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Ίσως υπάρχουν δύο θέματα τα οποία με απασχολούν ιδιαίτερα. Το πρώτο αφορά το δικαίωμα ασύλου και διεθνούς προστασίας. Διάβασα εντάχει την έκθεση αυτή, αλλά υπάρχει μεγάλη απεσιοδοξία ή σκεπτικισμός σε σχέση με το κοινό καθεστώς ασύλου για το 2012 ως προς το περιεχόμενό του πέρα από την προθεσμία. Επίσης, ε, εντάχει, θα ήθελα να σας μιλήσω για το καθεστώς και τις συνθήκες υποδοχής. Ποια είναι η διεθνής προστασία, το καθεστώς που προβλέπετε, γιατί υπήρξε μεγάλη κρίση σε κράτη-μέλη, όπως τη Γαλλία και το Βέλγιο το χειμώνα, μια ε, προβλεπόμενη κρίση η οποία όμως ε, είχε αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με την διεθνή προστασία. Άρα θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει μια κατάσταση αντιμετώπισης ε, κατεπηγουσών αναγκών. Τι γίνεται τη στιγμή που υπάρχει αίτημα διεθνούς προστασίας. Ένα άλλο θέμα αφορά την οικογένεια και το δικαίωμα διαβίωσης, με συγχωρείτε, της οικογένειας, της κοινή οικογενειακής ζωής. Ως προς την ένωση των οικογενειών, τι θα γίνει σε σχέση με την επανένωση των οικογενειών στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να μας πείτε πώς, έχει το, πώς προωθούνται αυτά τα οικογενειακά δικαιώματα, πώς θα γίνει με την ε, οικο, οικογενειακή επανένωση, τι προβλέπετε σε αυτό το καθεστώς. Η κυρία Γιάροκα. First of all, uh, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε τους τελευταίους ε, δέκα μήνες. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έμαθε πολλά από τις εκθέσεις και την ε, περσινή, την ετήσια, ιδιαίτερα σε σχέση με την κατάσταση των ε, Ρωμά. Θα ήθελα να εμβαθύνετε την κατάσταση σε σχέση με το έγκλημα, ναρκωτικά και άλλα θέματα που αφορούν την παραβίαση των δικαιωμάτων, ιδιαίτερα ως προς τα μικρά παιδιά των Ρωμά. Θα θέλαμε να τεθεί σε εφαρμογή πολύ σωστότερα, σωστότερα κατά το δυνατόν η οδηγία. Πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα σε τοπικό επίπεδο έτσι ώστε οι άνθρωποι να ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, να μπορούν να προσφύγουν όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους και πώς μπορούν να συνεισφέρουν έτσι ώστε να μάθουν πολύ καλύτερα για τα επίπεδα διακρίσεων σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν πιο ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Και ένα άλλο θέμα που θίξατε, όταν μιλάμε για την οικονομική συνεισφορά σε περιφερειακό επίπεδο και την εποπτεία ως προς τη, ως προς συλλογή στοιχείων για τη στρατηγική υπέρ των Ρωμά, πώς θα έχετε μια σωστή εικόνα, διότι όπως είπε και η κυρία Ζαουνακόβα, τους τελευταίους ε, δέκα μήνες είδαμε ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και ο χάρτης αντιμετώπισης των κρίσεων απαιτεί αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορέσετε να βοηθήσετε τα εθνικά προγράμματα δράσης προς αυτή την κατεύθυνση από την ε, πρώτη φάση του προγραμματισμού. Έχουμε τα σωστά στοιχεία. Η κυρία Κέλλερ. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά θα προσπαθήσω κάπως να περιοριστώ. Θα αρχίσω από τις ευκολότερες σε σχέση με την, οριζο... με την, οδηγία, την οριζόντια οδηγία ίσης μεταχείρισης σε σχέση δηλαδή και με τα θέματα που αφορούν περιπτώσεις αναπηρίας μέσα στα πλαίσια της, ε, του Οργανισμού Θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πώς εξελίσσεται, πώς έχει εξέλιξη αυτή της ε, οδηγίας στο Συμβούλιο. Δεύτερον, θα εγκρίνεται μία προσέγγιση αναχώρα για την επόμενη ετήσια έκθεση. Κρίνεται και αυτή η προσέγγιση είναι χρήσιμη. Επίσης έχετε δίκτες, έχετε συλλέξει δίκτες για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να ε, είναι πιο αποτελεσματική. Γενικότερα, στην επισκόπησή σας αναφέρετε ποιες χώρες καταδικάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και φαίνεται ότι η Ρουμανία βρίσκεται πρώτη στη λίστα με 135 υποθέσεις που εκκρεμούν. Γιατί υπάρχει τέτοια, ε, τέτοια, τόσο πολλές εκρεμείς υποθέσεις κατά ορισμένων συγκεκριμένα κράτων μελών. Επίσης, ποιες είναι οι πιο επίγουσες περιπτώσεις όπου θα πρέπει να αντιδράσετε, όπου θα πρέπει να αντιμετωπίσετε άμεσα. Ποιες είναι οι περιπτώσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τάχιστα κατά την άποψή σας. Ο κύριος Φως. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρώτη παρατήρηση, μάλλον ερώτηση, προς την ίδια κατεύθυνση με την κυρία Κέλλερ. Συχνά έχουμε μεμονωμένα προβλήματα και όταν συζητούμε αυτά τα μεμονωμένα προβλήματα έχουμε την εντύπωση ότι δεν είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο ή που θα μπορούσε να είναι ικανοποιητικό το επίπεδο. Γι' αυτό θα με ενδιέφερε πάρα πολύ. Βέβαια γνωρίζω ότι σε μια προφορική παρουσίαση δεν μπορεί κανείς να μας δείξει τι γίνεται και πώς αξιολογείται το κάθε τι, αλλά γενικά μια εκτίμηση θα παρακαλούσα. Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι καταρχήν με την κατάσταση στην Ευρώπη ή μήπως είμαστε στο μέσο όρο ή στη μετριότητα ή κάτω του μετρίου, ξέρω εγώ, μια γενική αξιολόγηση θα μπορούσατε να μας κάνετε. Θα ήταν πολύ ωφέλιμη, πολύ χρήσιμη. Μπορείτε να μας πείτε, είμαστε γενικά ικανοποιημένοι με κάποια μικροπροβλήματα, είμαστε γενικά ε, αρνητικοί. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων γενικά, και οι πολίτες ερμηνεύουν πολύ περισσότερα από αυτά που υπόσχεται ο χάρτης στην εφαρμογή του. Δεν θα πρέπει να κοιτάμε και να παρακολουθούμε και το περιεχόμενο του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εμένα πάντα κάτι μου λείπει από εκεί που το συζητάμε εδώ και χρόνια και είναι στην επικαιρότητα, η όλη κατάσταση στην Ισπανία με το νόμο περί προστασίας ε, των ακτών. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσμικά όργανα αφήνουμε στα κρύα του λουτρού ανθρώπους που τους απαλωτριώνουν και τους παίρνουν τις περιουσίες ε, δεν ξέρω βεβαίως αν θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε την ελευθερία της κυκλοφορίας των κεφαλαίων ή άλλη κινητικότητα. Τους αφήνουμε όλους στη μοίρα τους χωρίς να κάνουμε τίποτα και δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και τώρα απλώς διέτρεξα την έκθεση. Δεν το διάβασα. Αλλά θα πρέπει κάπου να το στιγματίσουμε. Εντάξει, εμένα δεν, με στεναχωρεί η ίδια η... Ε, απαλωτρίωση ή η δίμευση των περιουσιών. Ε, καλό αυτό, αλλά χρειάζεται και αποζημίωση. Δεν είναι ηθικά σωστό, δεν είναι πολιτικά σωστό και θα πρέπει να το πούμε. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι εκείνοι οι πολίτες που τους παίρνουν την περιουσία και δεν τους αποζημιώνουν και τρέχουν και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά μέχρι να δικαιωθούν ή να βγει απόφαση μπορεί να χρειαστούν και 15 και 20 χρόνια και πολλοί έχουν αποβιώσει και δεν το ζουν αυτό πια. Αφήστε δε που δεν είναι πάντα οι πολίτες όλοι ενήμεροι για τη ε, νομική οδό που μπορούν να ακολουθήσουν. Για να μην έχουν την αίσθηση οι άνθρωποι αυτοί ότι τους έχουμε εγκαταλείψει τη μοίρα τους. Ο κύριος Σταβάρες έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κέρον για την παρουσίαση αυτή. Θα ήθελα να αρχίσω με ένα στοιχείο που μας έδωσε η κυρία Ρέντινγκ που είπε ότι το ίμιση των προσφυγών των πολιτών δεν αποτελούν ε, αναπόσπαστο τμήμα της ε, κοινοτικής δικαιοδοσίας. Ίσως ε, δεν γνωρίζουν οι πολίτες τι είναι αρμοδιότητα της Ένωσης και τι των κρατών μελών ενδεχομένως ή αυτό δείχνει η έλλειψη ικανοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης που παπειλούνται τα δικαιώματα των πολιτών και αντιμετωπίζουν τους οργανισμούς αυτούς, όπως τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ως εγγυητές των δικαιωμάτων τους. Όταν δηλαδή υπάρχει αυτή η γενικότερη ε, απειλή θα πρέπει να διαδραματίσουν οι οργανισμοί έναν επιπρόσθετο ρόλο η συνάδελφος Κέλλερ μίλησε για την ε, σύνταξη της έκθεσης, εν μέρη τουλάχιστον αναχώρα, διότι ε, οι πολίτες θέλουν να βλέπουν πώς έχει η κατάσταση στη δική τους χώρα, δηλαδή πώς κατονομάζεται και ποιο είναι το καθεστώς της ισχύει στη δική τους χώρα. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η εντολή των πολιτών, αν θέλετε, είναι πολύ ευρύτερη από ό,τι προβλέπεται από τις συνθήκες και πιστεύω ότι η οργάνωση θεμελιωδών δικαιωμάτων αντιμετωπίζει αυτό το, αυτή την εντολή στρίκτο σένσου κάτι το οποίο ίσως δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστή ερμηνεία των συνθήκων και ιδιαίτερα της συνθήκης της Λισαβόνας. Ίσως η εντολή αυτή δηλαδή θα πρέπει να είναι πιο διευρυμένη για να λάβουν υπόψη και θέματα ελευθεροτυπίας και ελευθερίας του εκφράζεστε. Ιδιαίτερα ως προς τον ρόλο των ΜΜΕ. Αυτό μας απασχόλησε ιδιαίτερα στην Ουγγαρία και ίσως είναι προηγούμενο για άλλες χώρες. Δεν είναι θέματα εθνικής κυριαρχίας που αφορά την Ουγγαρία αποκλειστικά. Υπάρχει ένας κίνδυνος να απειληθούν τα δικαιώματα των, ανθρώπων και, των πολιτών και σε άλλες χώρες. Το ίδιο αφορά και την ομοφιλοφοβία σε χώρες που αντιμετωπίζουν πιο οξύ πρόβλημα. Θα θέλαμε η οργάνωση θεμελιωδών δικαιωμάτων να ε, δρά πιο άμεσα και με μεγαλύτερη πεποίθηση. Αυτό είναι ύψη της σημασίας, γιατί θα πρέπει να φτάσουμε σε μια φάση, να φτάσετε μάλλον, σε μια φάση ορίμανσης η έκθεση είναι άκρος ενδιαφέρουσα, θα πρέπει να αναγνωστεί με προσοχή, αλλά φαίνεται σαν να βρισκόσαστε σε διερευνητική φάση, ενώ υπάρχουν απτές παραβιάσεις δικαιωμάτων που θα πρέπει να στυλιτεύονται καλύτερα ή περισσότερο από τις εκθέσεις, δηλαδή ε, πολλές φορές χώρες αναφέρουν ότι βρίσκονται σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτή που κατονομάζει η οργάνωση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό πιστεύω ότι η εντολή θα πρέπει να διευρυνθεί ή να μην ερμηνεύεται συσταλτικά αλλά διασταλτικά, όπως είδαμε στην περίπτωση των ΜΜΕ στην Ουγγαρία. γιατί δεν βλέπω να ε, στυλιτεύεται ιδιαίτερα τις περιπτώσεις παραβίασης του δικαιώματος του εκφράζεστε. Ο κύριος Κλέης έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Στην ετήσια έκθεση, στο κεφάλαιο 7, γίνεται λόγος για τη συμμετοχή πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης. Και μεταξύ αυτό γίνεται λόγος και για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, για την πρωτοβουλία πολιτών κτλ. Πουθενά όμως δεν γίνεται λόγος για την κατάσταση ε, της ελευθερίας της έκφρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλά κράτη-μέλη. Που, ενώ η ελευθερία της έκφρασης είναι από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και χωρίς αυτό δεν νοείται η δημοκρατία. Διαπιστώνουμε όμως ότι σε πολλά κράτη-μέλη το δικαίωμα της ελευθερίας στην έκφραση καταστέλλεται όλο και περισσότερο. Και κατά παράδοξο τρόπο αυτό γίνεται υπό το πέπλο της καταπολέμησης του ρατσισμού ή του λεγόμενου ρατσισμού. Σε κάποια κράτη-μέλη κατεβάλλονται προσπάθειες έτσι ώστε κάθε συζήτηση, κάθε αντιπαράθεση ε, για θέματα ένταξης και μετανάστευσης να ε, είναι αδύνατη. Το καλύτερο παράδειγμα είναι οι κάτω χώρες, όπου ένας ηγέτης κόμματος, ο Χέρτ Wilders, αυτή τη στιγμή είναι στα δικαστήρια και κατηγορείται και ε, κινδυνεύει να καταδικαστεί για διακρίσεις, για υποδάβληση του μίσους, του ρατσισμού κτλ. Μα τι έκανε ε, τόλμησε να αμφισβητήσει μια πολιτική που κανονικά είναι καθήκον κάθε εκλεγμένου βουλευτή. Λοιπόν, ο οργανισμός σας θεωρεί την ελευθερία της έκφρασης πυλώνα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μπορούμε στο μέλλον να περιμένουμε ε, να λάβει ε, σαφή και μονοσήμαντη θέση ο οργανισμός υπέρ αυτής της ελευθερίας και κατά ε, της κατάχρησης που γίνεται αυτών των μεγάλων ε, ιδεοδών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης του ρατσισμού για να καταστέλλεται και να φημώνεται κάθε συζήτηση. Ευχαριστώ. Επανέρχομαστε τώρα στους εκπροσώπους ε, του οργανισμού, ίσως με την ίδια σειρά ή την αντίστροφη, όπως θέλετε. Ο κύριος Κέρουμ πρώτος, για να απαντήσει σε ερωτήσεις που έγιναν. Thank Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα χαρά μου να έρχομαι εδώ και να ακούω τόσο <laughs> πολλές περίπλοκες ερωτήσεις, σχόλια που εμπλουτίζουν ε, την εργασία μας και ακριβώς αυτά όλα προωθούν τα θέματα. Θα ήθελα να απαντήσω στις περισσότερες ερωτήσεις και μετά θα μοιραστούμε τις απαντήσεις ε, με την κυρία Μπραντ Έγινε μια πρώτη ερώτηση, αλλά αναφερθήκατε και άλλοι σε αυτό, είναι στο θέμα του ασύλου και στην προστασία προσφύγων στην Ευρώπη σήμερα. Μάλιστα αναφερθήκατε ρητά και στην κατάσταση στα σύνορα της Ελλάδας που υφίσταται μεγάλη πίεση, κατακλείζεται η χώρα είναι πολύ σημαντικό όταν συζητούμε για αυτά τα θέματα να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Είναι πολλές οι κρίσεις των προσφύγων, ας πούμε, παντού στον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γενικά το κατατάσσουμε αυτό σε θέματα ανθρωπιστικής κρίσης. Και έχουμε πολλά προβλήματα ανθρωπιστικής κατάστασης που δεν έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μπορεί να είναι δραματικά και χρειάζονται αντιμετώπιση, αλλά δεν είναι θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτά. Ε, ούτε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, αυτό που βλέπουμε τώρα ε, και λέμε στην έκθεσή μας και έχουμε τακμηριώσει και είναι έτσι μοναδικό είναι η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις ανθρωπιστικές κρίσεις. Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Όπως σας είπα, η κατάσταση στα κέντρα κράτησης ποια είναι και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση εδώ και κάπως ο καιρό. Επίσης δεν υπάρχει και πρόσβαση. Κάνεις στις διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Να εξετάζονται οι περιπτώσεις, οι υποθέσεις του καθενός χωριστά. δυστυχώς ε, σήμερα παραμένει η κατάσταση εξίσου έκτακτη και κατεπίγουσα όπως και πριν από μερικούς μήνες που καταθέσαμε την έκθεσή μας μετά από έρευνα που είχαμε κάνει επί τόπου αρχές του 2010. Για τις μονάδες Rabbit της Frontex έχουμε την αίσθηση και την εντύπωση, βέβαια χωρίς να είναι η βασική μας εστίαση, πάντως αποκομίσαμε την εντύπωση από τη μελέτη ότι η Frontex διαδραματίζει ρόλο κλειδί στην προστασία των ε, δικαιωμάτων των προσώπων αυτών ε, να ε, τη χάνουν υποδοχής στα σύνορα και μετά να διαβιβάζονται, να, να μεταφέρονται στις αρμόδιες αρχές. Μπορούμε, θέλετε, να συζητήσουμε την εντολή της Frontex, αλλά στα πλαίσια της εντολής νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά και προστατεύει τα δικαιώματα των προσώπων που φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τον καιρό το εξετάζουμε σε μεγαλύτερο βάθος αυτό το θέμα. Στα πλαίσια της μελέτης και της εξέτασης των εξωτερικών συνόρων και στη Μεσόγειο, στα θαλάσσια σύνορα, σε τρία αεροδρόμια και ε, σε κάποια χερσαία σύνορα για να δούμε κατά ξηρά θάλασσα και αέρα τι γίνεται ε, στα σημεία εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορούμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις αυτές. Ίσως του χρόνου, ας ελπίσουμε μάλλον του χρόνου, να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε εκτενέστερα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Για την οδηγία επαναπροώθησης και πάλι θα την ενημερώσουμε. Εγώ δεν έχω τα πιο πρόσφατα στοιχεία στη διάθεσή μου εδώ, αλλά θα είναι ένα από τα σημεία που θα χρειαστούν ενημέρωση στην επόμενη τήσια έκθεση και στις μελλοντικέ. Από τις έρευνες που κάνουμε γενικά και τις μελέτες εκεί, γιατί έχουμε μια εμπειρία και ένα ρυθμό ήδη εκθέσεων για το άσυλο και την υποδοχή ε, ατόμων που ζητούν άσυλο ή παιδιών, ε, συνόδευτων ε, ανηλίκων, τι διαπιστώνουμε, ότι χρειάζεται περισσότερη συνεργασία, συντονισμός In order to, as I said... μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σας είπα και προηγουμένως και ο συντονισμός και η αλληλεγγύη θα πρέπει να θεωρείται ως αναπόσπαστο τμήμα της προστασίας και του καθεστώτος προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτά είναι εξάλλου διδάγματα που έχουν εξαχθεί από την περίοδο ε, των προσφύγων από την Ινδοκίνα στο τέλη της δεκαετίας του 70 που ε, αναζητούσαν διεθνή προστασία. Αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν να διαφυλαχθούν τα ε, δικαιώματά τους. Έχουμε λοιπόν εξαγεί πολλά ε, συμπεράσματα και διδάγματα από εκείνη την περίοδο που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, στην επανένωση των οικογενειών. Γνωρίζουμε ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν δοκιμάσει διάφορα μοντέλα περιορισμού. Ε, της επανένωσης των οικογενειών και της οικογενειακής ζωής. Υπάρχουν και υποθέσεις στο Στρασβούργο που εκκρεμούν στο δικαστήριο για να διαπιστωθεί ε, πού βρίσκονται ακριβώς τα όρια, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα ε, στο δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή που είναι και το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από την άλλη να αποφασίσουμε ποιος έχει δικαίωμα ε, να παραμένει στην επικράτεια ενός συγκεκριμένου κυρίαρχου κράτους. είναι λεπτές ισορροπίες εδώ, ξέρετε, και Ε, περιμένω κι εγώ με μεγάλη περιέργεια να δω πού θα τραβήξουν αυτή τη διαχωριστική γραμμή. Τι άλλο. asylum. Ε, ε, I think that was, uh, Then that, uh, Στη συνέχεια. Γενικότερα, Δεν θυμάμαι ποιος ρώτησε, η κυρία Σδάνοκα. Αν ε, ο ρόλος μας έχει αναχθεί, έχει περιοριστεί στη σύνταξη εκθέσεων και στη διοργάνωση συνεδριάσεων. Ε, όχι. Ε, έχουμε μεγαλύτερο έργο από αυτό. Συλλέγουμε στοιχεία που θα πρέπει να δίνουμε στα ευρωπαϊκά κράτη και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με παροχή συμβουλών αλλά να βασίζονται πάντα σε στοιχεία. Και προφανώς είναι η δουλειά μας να συλλέγουμε στοιχεία είτε δευτερογενή και πρωτογενή αν δεν υπάρχουν. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή Όλος ο κλάδος αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, είναι δουλειά μας να μεταφέρεται στην πράξη, να ξεφεύγει από την αόριστη θεωρία και να γίνεται καθημερινή δουλειά. Ε, αλλά, όπως είπε και ο πρόεδρος και η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μας, έχουμε απαντήσει σε αιτήματα του Κοινοβουλίου ε, για... την Ευρωπαϊκή Εντολή Ερεύνηση για τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών, το PNR, δύο φορές δηλαδή, Είναι πολλαπλή η εντολή μας και η αποστολή μας, αλλά είναι κλειδί αυτό και βασικό η παροχή στοιχείων και ε, συμβουλές με τεκμηρίωση ακριβώς με βάση στατιστικά στοιχεία. Για τους Ρωμά, βεβαίως θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακόμα περισσότερο, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και έχουμε δεσμευτεί. Το 2010 τι έγινε. Αυτό το θέμα ήρθε στο κέντρο το, της υπόθεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την περιφέρεια που ήταν στο παρελθόν και θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ περισσότερο στις προκλήσεις. Και εδώ η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ε, σημαντικό βήμα πρόοδου στην κατεύθυνση αυτή. Είναι πολλές ελπιδοφόρες εξελίξεις. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, αλλά ελπίζω να το προωθήσουμε. Κάτι που θα κάνουμε μαζί σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Παγκόσμια Τράπεζα θα κάνουμε ε, μια μεγάλη έρευνα στα νοικοκυριά. Για να δούμε ε, πώς συνεργάζονται και ποια είναι η σχέση των τοπικών, των τόπιων πληθυσμών και ε, με τους ε, ντόπιου Ρωμά και πού είναι θέμα ε, διάκρισης και πού υπάρχουν άλλα προβλήματα και ζητήματα απλής ένδυας εντός εισαγωγικών το απλής. χρειάζεται περισσότερο να ερευνήσουμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει για να έχουμε μια στοχευμένη ε, παρέμβαση και σωστή. Ένα από τα στοιχεία που ρωτήσατε επίσης είναι η συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων που έχουν ε, οι κοινότητες αυτές. Είχαμε πολλές συζητήσεις με ε, φορείς των κρατών μελών για θέματα ισότητας και δικαιωμάτων. Γιατί στη μεγάλη έρευνα που κάναμε αποκαλύψαμε ότι πολλά από τα θύματα των διακρίσεων δεν ξέραν πού να αποτανθούν για τα δικαιώματά τους. Τώρα υπάρχουν ε, φορείς ισότητας και στα 27 κράτη-μέλη. Ε, θα πρέπει ε, να ενημερώνονται οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί, ομάδες ομάδες ατόμων στις κοινωνίες για την ύπαρξη. Αφού έχει στηθεί η δομή, αλλά θα πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος ότι υπάρχει και μπορεί να απευθύνεται εκεί. Γίνονται πολλές σημαντικές συζητήσεις μεταξύ αυτών των φορέων Μερικοί εργάζονται πολύ καλά, ας ε, διδαχθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο κι εμείς. Ε, και υπογραμμίζεται επίσης και στην ανακοίνωση ότι βοηθούμε τα κράτη-μέλη για τις εθνικές τους στρατηγικές, βέβαια πρώτα απ' όλα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επί σειρά ετών είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για ε, κοινή διακυβέρνηση, για συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες. Υπάρχουν πολλά ζητήματα εκεί και προκλήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τους Ρωμά. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η προσπάθεια, έτσι, δέσμη μέτρων και με χαρά να συνεχίσουμε να τους συζητούμε και με το Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή σας επόμενους μήνες. Για την οριζόντια οδηγία Κυρία Κέλλερ. Έφυγε. Α, δεν πειράζει. Πολύ από τη δουλειά που κάνουμε, οι μελέτες και οι έρευνες για την αναπηρία οι ε, κάποιες άλλες μελέτες για την καταπολέμηση ε, της ομοφιλοφιλοφοβίας Ε, χρειάζεται ακριβώς αυτή η εγκάρση οριζόντια οδηγία. Ελπίζω να χρησιμοποιείτε για την προώθηση της θέσης ισχύ της οδηγίας αυτής. Θα συνεχίσουμε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή, αν υπάρχουν ιδιαίτεροι τομείς που ε, σας ενδιαφέρουν ε, περισσότερο, παρακαλώ μας το δηλώσετε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κάτι άλλο που ρώτησε η κυρία Κέλλερ, πόσο χρήσιμοι είναι οι δείκτες. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο αυτό το πεδίο. Αλλά οι δείκτες μας βοηθούν ακριβώς να επικεντρωνόμαστε σε κάποιους στόχους και να μετράμε την πρόοδο που έχει γίνει. Παντού, σε όλου του τομείς, όχι μόνο στα θεμελιώδη δικαιώματα και στην οικονομία, σε πολλούς κλάδους που έχουμε δείκτες, είναι χρήσιμοι και σε εμά. Και το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και το προωθούμε. Ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα στην Ευρώπη. είναι δύσκολο ε, να αυτό, προσδιορίσεις αυτό, γιατί ο καθένας που υφίσταται μια διάκριση έχει πρόβλημα με τα δικό του δικαίωμα, το θεωρεί το σημαντικότερο. Πάντως θα τολμούσα να πω ότι η κατάσταση στα σύνορα, όπως τα συμπεριέγραψα, είναι από τις ε, πιο σημαντικές υποθέσεις που πρέπει να λυθούν Βεβαίω το θέμα το Ρωμά είναι πάρα πολύ σημαντικό και κεντρικό και κομβικό, αλλά ε, χρειάζεται ανάπτυξη μακροπρόθεσμη λύση. Ενώ αυτό που παρατηρούμε στα ε, σύνορα, στα κέντρα κράτησης, είναι στα χέρια μας να το αλλάξουμε. Και εκεί περιπλέκονται πολύ τα πράγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μπορούμε να τα αλλάξουμε. Uh, Κύριε Βος, ρωτήστε αν είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση στην Ευρώπη γενικά. Νομίζω ότι η Ευρώπη είναι κατεξοχήν ε, η περιοχή του κόσμου με τον υψηλότερο βαθμό γνώσης και ευαισθητοποίησης ό,τι αφορά τα θέματα θεμελιδών δικαιωμάτων για τη διακριτική μεταχείριση. Νομίζω ότι προχωρήσαμε πολύ ό,τι αφορά αυτή την ίση μεταχείριση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση, έχουμε πολλούς αρμόδιους φορείς και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Φυσικά μας απομένουν πολλές προκλήσεις, κάτι που φάνηκε και στην ετήσια μας έκθεση τη φετινή. Ναι, μεν είμαι αισιόδοξο από την άποψη ότι υπάρχει συνειδητοποίηση και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζουμε το θέμα αυτό Ταυτόχρονα όμως μας απομένουν πολλές προκλήσεις. σημείωσε πάντως το ζήτημα που επισημάνατε για τα δικαιώματα ε, της γης και θα το ελέγξω περαιτέρω και το θέμα των δημεύσεων περιουσιών κτλ. Ο κύριος Σταβάρες αναφέρθηκε στην εντολή του οργανισμού. Αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Τι είδου ε, οργανισμό θέλουν τα κρατημέλη μελη Κομισιόν, το Συμβούλιο για το μέλλον. Εμείς ε, δεν διστάζουμε να υπογραμμίσουμε ορισμένα ζητήματα και να θίξουμε τα κακό σκήμενα στην ετήσια έκθεσή μας. Εσείς είπατε να συντάξουμε έκθεση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη σχετική νομοθεσία στην Ουγγαρία. Για μια συγκεκριμένη πάντως πριν από μερικά χρόνια, πέρυσι αν δεν κάνω λάθος, μας είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να αποφαθούμε σε ό,τι αφορά το, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στη Λιθουανία και να συντάξουμε σχετική έκθεση. Αλλά δεν μπορούμε να συντάξουμε ειδική έκθεση για μια συγκεκριμένη χώρα. Απλώ εκπονήσαμε μια έκθεση με την κατάσταση σε έξι χώρες και την παρουσίαση της αντίστοιχης νομοθεσίας σε έξι χώρες. Από αυτή την άποψη, ίσως μια-δυο χώρες ξεχωρίσουν ως πιο αδύναμες ό,τι αφορά αυτή την κατάσταση. Πάντως, εξατομικευμένη έκθεση για μια χώρα σίγουρα έχει περισσότερο βάρος από μια συγκριτική μελέτη αλλά ε, μέχρι στιγμής με την εντολή μας όπως έχει διαμορφωθεί αυτό προβλέπεται. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία έκφρασης, έκφρασης και την αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας έκθεσης και της, έκφρασης και της αποφυγής δηλώσεων μυσαλλοδοξίας ή υποκίνησης μίσους κτλ. Αυτή είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία που επιδιώκουμε να την αναζητούμε και είναι κάτι που μας ενδιαφέρει επίσης. Αυτά. Κυρία Κέρις, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε. Ευτυχώς ο, ο Μάρτιν κάλυψε σχεδόν τα πάντα και βλέπω ότι έχουμε ξεπεράσει και την ώρα μας. Γι' αυτό είναι ευτυχή συγκυρία που εγώ δεν χρειάζεται να μιλήσω πολύ. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία έκφρασης, επανέρχομαστε και πάλι στο ζήτημα του πολιετούς πλαισίου. Δεν είναι, το θέμα της ελευθερίας έκφρασης δεν είναι κάτι αυτοτελές και αυτόνομο. Το εξετάζουμε πάντα σε συνδυασμό με άλλα θέματα. Ή το θέμα της υποκίνησης του μίσους, με μισαλόδοξες δηλώσεις κτλ. Όταν υπάρχουν μεμονωμένες παραβιάσεις, υπάρχουν αρμόδιοι φορείς που μπορούν να ελέγξουν τέτοιες καταγγελίες, αλλά δεν εμπίπτει αυτό στη δική μας εντολή να συγκεντρώνουμε τέτοιες καταγγελίες. Υπάρχουν αρμόδια όργανα που μπορούν να τις εξετάζουν. Σε ό,τι αφορά το τοπικό επίπεδο και τους δείκτες, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το έργο που έχει γίνει σε ό,τι αφορά την ε, συγκέντρωση δικτών από πολλούς φορείς και εμείς συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια εκπόνησης δικτών. Και φυσικά προσπαθούμε να συνδέσουμε αυτό το ζήτημα με τους τοπικούς ε, φορείς, γιατί οι τοπικοί φορείς, τα τοπικά δίκτυα συνεργασίας εκδήλωσαν ενδιαφέρον για αξιοποίηση και της δική μας ε, εμπειρίας. Θέλουμε φυσικά αυτό το θέμα να φτάσει, να κατέβει στο τοπικό επίπεδο, όπως είπε η κυρία Γιάρουκα. Και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Ό,τι αφορά το τελευταίο θέμα για την ηθαγένεια, η υπηκότητα ή τους απάτριδες, το μεγάλο τους αριθμό στις βαλτικές χώρες, αλλά δεν είναι μόνο οι βαλτικές χώρες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα του νομικού καθεστώτος και Όντως αυτό που επισημάνατε μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε τη συμμετοχή τουλάχιστον σε ευρωεκλογέ. Γιατί όντως αυτό το θέμα της συμμετοχής, ε, της δυνατότητας ε, για ψήφους σε ευρωεκλογέ εμπίπτει στο κεφάλαιο αυτό. Ίσως <clears throat> θα, μπορούμε, θα μπορούσαμε με τη συγκέντρωση των στοιχείων να κάνουμε εμείς μια τέτοια έρευνα, γιατί δεν συγκεντρώνουν τέτοια στοιχεία τα κράτη-μέλη, αλλά αν μπορέσουμε τέτοια στοιχεία να τα συμπεριλάβουμε στο κατάλογο, για, στο κεφάλαιο για την ηθαγένεια, προκειμένου να ενισχύσουμε αυτό το κεφάλαιο για την ηθαγένεια, γιατί μέχρι στιγμής αυτά τα θέματα δεν βρέθηκαν στο επίκεντρο τη δική μα προσοχή, αλλά αν επεκτείνουμε αυτό το κεφάλαιο με τέτοια ζητήματα θα ήταν ενδιαφέρον. Θα μπορούσε κάλλιστα να βρουν τη θέση του σε αυτό το κεφάλαιο για την ηθαγένεια. Εσείς είπατε ότι αυτή η κατάσταση των απάτριδων, αλλά και η πρόσβαση στην υπηκότητα είναι κάτι που δεν εμπίπτει ούτε και αυτό στην εντολή της, ούτε του οργανισμού, ούτε καν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά όμως την συμμετοχή στις εκλογές, αυτό μας ενδιαφέρει. Θέλουμε ουσιαστική συμμετοχή όλων των πολιτών, των κατοίκων και αυτό θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε σε μελλοντικά προγράμματα. Και επανέρχομαι στα τελικά συμπεράσματα, βέβαια τα λιγότερο ευχάριστα αφορούν τους περιορισμούς και τις αδυναμίες. Και επανέρχομαι στο πρώτο ζήτημα και των μελλοντικών συζητήσεων, που αφορά το θεματολογικό πλαίσιο του οργανισμού για τα επόμενα χρόνια. Και όλοι οι ενδιαφερόμενοι αλλά κυρίως οι ηθήνοντες, που, λαμβάνουν τις αποφάσεις, ενδιαφέρονται ε, για το θέμα αυτό και όντως ε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα θέματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως να συμπεριληφθούν στις συζητήσεις ή να συμπεριληφθούν στις διαπραγματεύσεις. Και εμείς περιμένουμε την έκβασή τους για να δούμε σε ποια θεματολογία θα επικεντρωθούμε. Σας ευχαριστώ. Προς το παρόν σταματάμε εδώ τη συζήτηση. Κάποιος ζήτησε το λόγο για συμπληρωματικό σχόλιο, αλλά σας υπενθυμίζω ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω στο πρόγραμμά μας. Οπότε αν έχετε παρατηρήσει παρακαλώ τηλεγραφικά. Ναι, εμείς ζητήσαμε έκθεση για το νόμο, τον Ουγγρικό νόμο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά μας είπατε ότι ο οργανισμός δεν ασχολείται με μεμονωμένες χώρες. Ζητήσαμε όμως και συγκριτική μελέτη για την ελευθεροτυπία, για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε όλες τις χώρες μελέτη. Κάτι που είναι τελείως διαφορετικό. Ο κύριος Κέρομ. Όντως, το Κοινοβούλιο έθεσε τέτοια αίτηση και είπαμε ότι με την ισχύουσα εντολή του οργανισμού, αλλά και με βάση τους σπόρους μας θα ήταν αδύνατον να καταρτήσουμε τέτοια έκθεση. Φυσικά κάθε έτοιμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα και το αναλύουμε διεξοδικά, αλλά ούτε και αυτή τη φορά είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίμα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κέρουμ, τον Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας και θα πρέπει τώρα να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα σημεία της ημερήσης διάταξης. We got some minutes. Έχουμε μείνει λίγο πίσω, όπω είπα. Έχουμε ολιγόλεπτη καθυστέρηση σε σχέση με το πρόγραμμα και περνάμε στο σημείο 5 που αφορά την συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία τη Ισλανδία και του Βασιλείου τη Νορβηγία για τη διαδικασία παράδοση μεταξύ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των δύο χωρών, Ισλανδία και Νορβηγία δηλαδή. Θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεση που εκπώνησε ο συνάδελφό μα, Ρούι ταβάρε ο εισηγητής της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Μην ξεχνάτε ότι το 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνένεσε στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας για την αμοιβαία δικαστική αρρωγή σε ποινικά θέματα. Τώρα ασχολούμαστε με μια άλλη διεθνή συμφωνία που συνήθεια αυτή τη στιγμή που συνήθως τη φορά μεταξύ Νορβηγίας και Ισλανδίας. Αφορά τη διαδικασία παράδοσης και στόχο έχει να εφαρμόσει μεταξύ των ενωσιακών χωρών μελών και της Νορβηγίας και της Ισλανδίας τις ίδιες αρχές που διέπουν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τη σχετική διαδικασία. Μια παράλληλη διαδικασία αφορά τη συμφωνία που συνήθε με την Ορβηγία και την, ε, Ισλανδία για την αμοιβαία δικαστική αρρωγή σε ποινικά ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου εν ώψη της επίσημης ε, υιοθέτησης της συμφωνίας αυτής με βάση το άρθρο 218 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Άρθρο που προϋποθέτει τη συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας για να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του. Θα δώσω δηλαδή το λόγο στον κύριο Ταβάρες και μετά θα προσδιορίσουμε τη διορία για τις τροπολογίες. Κύριε Ταβάρας, έχετε το λόγο. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Well, Norway and Iceland, of course. Όπως ξέρετε, η Νορβηγία και η Ισλανδία αποτελούν μέρος του χώρου Σέγγεν και ε, εάν το, αν και το ε, Σέγγεν και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δεν συμπίπτουν, δεν συμπίπτουν απόλυτα, αλληλοσχετίζονται και γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσουν από κοινού και οι δύο χώρες θα ήθελαν να προσχωρήσουν στο καθεστώς του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης με βάση αυτή την κοινή διαδικασία παράδοσης μαζί με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως αναφέρει και, αναφέρεται και στην έκθεσή μου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αντιταχθούμε στο αίτημα αυτό. Δηλαδή να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο που ήδη προϋπάρχει για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δύο χώρες έχουν ε, πολύ ε, καλή γραφή ως προς την ε, μεταχείριση των φυλακισμένων, δεν υπάρχει θανατική ποινή και συμμετέχουν σε άλλες πτυχές της διαδικασίας της ασφάλειας, ελευθεριών και δικαιοσύνης. Άρα δεν υπάρχει βασική, κάποια βασική αντίρρηση έτσι ώστε να συμμετάσχουν στην διαδικασία παράδοσης. Υπάρχουν όμως ορισμένες λεπτομέρειες που μας απασχολούν. Καταρχήν για την άρση, το καθεστώς άρσης, έτσι ώστε να μην γίνεται παλήθευση του διπλού χαρακτήρα ως προς το ποινικό δίκαιο και την εγκληματικότητα και εδώ μιλάμε για το σοβαρό έγκλημα. Έγιναν λοιπόν συζητήσεις σε σχέση με τα αδικήματα που προβλέπονται ιδιαίτερα όταν πρόκειται για βοήθεια έτσι ώστε να παραμείνει ε, ο υπόδικος αυτός ή ο εγκληματίας στη χώρα. Ε, δηλαδή να αρθεί η εξέταση του διπλού χαρακτήρα ε, εγκληματικότητας, διότι έχει μεγάλη σημασία για ορισμένους πολίτες στην Ένωση να υπάρχει ένας τέτοιος έλεγχος που έχει ειδικό πολιτικό βάρος. Όμως υπάρχουν χώρες που δεν ε, ε, αποφασίζουν ως προς την άρση του ερευνητικού χαρακτήρα, του διπλού ερευνητικού χαρακτήρα για αδικήματα. Πολλές φορές ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, ιδιαίτερα όταν μιλήσαμε για το θέμα της, του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, όπως το συζητήσαμε στην τελευταία Ολομέλεια στο Στρασβούργο, δηλαδή ότι έχει αρκετά κενά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα ε, κριτήριο ε, ανθρωπισμού ως προς την εφαρμογή δηλαδή του ε, Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, δικαιώματα των υποδίκων, δικαιώματα των εναγωμένων, δικαίωμα μετάφρασης και διερμηνίας και ούτω καθεξής. Φυσικά δεν είναι τέλειο αυτό το μέσο, είναι ένα επικοδομητικό μέσο και δεν βλέπω το λόγο να αντιταχθούμε έτσι ώστε να προσχωρήσουν και η Νορβηγία και η Ισλανδία. Άρα, στο προσχέδιο που σας έχω υποβάλει, αυτό ακριβώς προτείνω. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνενέσει στη σύναψη συμφωνίας. Έχουμε προθεσμία μέχρι τις 20 Ιουνίου για υποβολή ε, τροπολογιών, αν δεν κάνω λάθος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ταβάρες, ήσασταν ιδιαίτερα συνοπτικός. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να λάβει το λόγο ούτε η Ουγγρική Προεδρία. Υπάρχουν ε, μέλη που θα ήθελαν να σχολιάσουν την ε, παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης του κυρίου Ταβάρες. Φαίνεται πως όχι, κανείς δεν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Εάν όχι, Απλώς ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών έχει οριστεί για τις 20 Ιουνίου. 20 Ιουνίου λοιπόν για την υποβολή τροπολογιών για την έκθεση αυτή του κυρίου Ταβάρες. Ωραία, θαυμάσια, κλείσαμε και με αυτό το θέμα και ε, φτάνουμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης σε σχέση με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και διαβίβαση στοιχείων από τους αερομεταφορείς των δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών PNR, προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα αυτό συζητήθηκε με επικεφαλή στην κυρία Ιντβελτ και θα πρέπει να εξετάσουμε τώρα την ε, σύσταση αυτή. Γι' αυτό δίνουμε το λόγο στην κυρία Ιντβέλτ να μας ενημερώσει για την ε, κατάσταση και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί ή μπορούν να αναλυφθούν από τις πολιτικές ομάδες σε σχέση με τη Συμφωνία PNR. Και θα ακούσουμε και την ε, Επιτροπή ή την Προεδρία. Ευχαριστώ, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομη, διότι δεν υπάρχει καμία πρόταση σύστασης, κανένα προσχέδιο σύστασης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε να συζητήσουμε και τίποτα. Εάν δεν παρακολουθήσετε το θέμα εκ του σύνεγγης, θα ήθελα να σας πω ότι έχει επέλθει συμφωνία με την Αυστραλία, η οποία ισχύει ε, προσωρινά σε σχέση με τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων, PNR. Εμείς ήμασταν πολύ επικριτικοί ως προς αυτές τις συμφωνίες και με τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας θα πρέπει να συνενέσουμε σε αυτή την προσωρινή συμφωνία με την Αυστραλία και επίσης με τις συμφωνίες με ΙΠΑ και Καναδά. Θα θυμόσαστε ότι πέρσι το Μάιο είχαμε αναστείλει αυτή την ε, ψηφοφορία για να κερδίσουμε χρόνο, έτσι ώστε να διαπραγματευτούμε μια καλύτερη συμφωνία. Ε, ε, πρόθεσε τη διαπραγμάτευση από κοινού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Αυστραλία για να συνενέσουμε και θεωρήσαμε ότι το Συμβούλιο θα ήταν ενδεχομένως σε θέση να λάβει μια απόφαση με βάση τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων την προηγούμενη εβδομάδα. Κάτι τέτοιο όμως δεν ίσχυσε δυστυχώς. Τα κράτη-μέλη έχουν επιφυλάξει αντιρρήσεις. Πολλές ε, σχετίζονται με το περιεχόμενο του προσχεδίου συμφωνίας, άλλες είναι τυπικές, ιδιαίτερα όταν υπάρχει καθεστώς αυτοεξαίρεσης για ορισμένες χώρες και θέλουν μία περίοδο περισυλλογής τριών μηνών για να δεχτούν αυτό το πλαίσιο. Το Συμβούλιο λοιπόν δεν έχει αποφανθεί και άρα δεν μπορούμε να προβούμε προς μια σύσταση. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε και τίποτα βεβαίως αυτό, διότι οι σκιώδεις, όλες οι πολιτικές ομάδες και εγώ από κοινού συνεργαζόμαστε όχι μόνο ως προς συμφωνία της Αυστραλίας αλλά και αυτές των, με τις ΗΠΑ και την, τον Καναδά. Θα ε, εξετάσουμε και το, καθεστώς, το ευρωπαϊκό καθεστώς PNR διαβίβασης προσωπικών δεδομένων των επιβατών. Γι' αυτό έχουμε μια προφορική ερώτηση για την Ολομέλεια του Ιουλίου, έτσι ώστε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο. Η Πολωνική Προεδρία θα είναι ιδιαίτερα δραστήρια επί του θέματος. Αυτό μας υποσχέθηκε. Σήμερα το πρωί το συζητήσαμε με τους σκιώδεις και αποφασίσαμε για ένα κοινό κείμενο και για διαδικαστικούς λόγους προθεσμίας και ούτω καθεξής. Η προφορική ερώτηση δεν θα είναι ερώτηση της ΛΥΜΠΕ, αλλά θα είναι μια κοινή προφορική ερώτηση όλων των πολιτικών ομάδων. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να προσθέσω κάτι για την ουσία του σχεδίου. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Αν θέλουν τα μέλη να σχολιάσουν, ή θέλουν επιπρόσθετα στοιχεία μπορούν να μου τα ζητήσουν. Ωραία λέει ο πρόεδρος, χωρίς μικρόφωνο. Thank you. Thank you, Η Επιτροπή εντάχει βεβαίως ε, θα ε, συζητηθεί το θέμα τον Ιούλιο και το προσμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον στην Ολομέλη. Short updating. Ε, ωραία. Θα υπάρχει ενημέρωση λοιπόν για, για το σχέδιο το οποίο δεν έχει ακόμα υπάρξει, δεν έχει ακόμα ανακύψει, το σχέδιο ε, σύστασης. Προχωράμε πολύ καλά. Πολύ καλά και πολύ γρήγορα στο επόμενο θέμα που είναι το υπαριθμόν 7 σε σχέση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για, ως προς την ετήσια έκθεση για το 2010 για την προστασία δεδομένων. Θα ακούσουμε την παρουσίαση του κυρίου Χαστίνγκς. Ε, προβλεπόταν για τις 11 η συζήτηση, ο κύριος Χάστινγκς ε, δεν είναι παρόν, άρα ας διακόψουμε με χρυσό του προσέλθει ο Πίτερ Χάστινγκς με την ομάδα του για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε από το να πάμε στο επόμενο σε σχέση με την ίση μεταχείριση προσώπων και ούτω κάθεξη. Γιατί ο Ραούλ Ρωμέβα θα βρίσκεται εδώ στις 11.30 άρα διακόπτουμε για μισή ώρα. Σας ευχαριστώ. Let's take a break. Okay. Gianni siamo stati fin troppo rapidi, potete venire un po' prima alle 11 meno un quarto? cioè fra, fra un quarto d'ora. Fra un quarto d'ora, eh. We've just, excuse me, if you, if you, if you allow me for a second, we just heard that they are on their way. Μου λένε, αν μου επιτρέπετε, ότι καταφθάνουν οι εκπρόσωποι ε, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο κύριος Χάστινγκς και ο κύριος Βουταρέλη. Οπότε το διάλειμμα κάντε το Τέταρτο παρακαλώ, όχι μισή ώρα. Στις παρατέταρτο θα συνεχίσουμε. Μα όλα τα μέλη έχουν υπολογίσει ότι η συζήτηση θα γίνει στις 11. Υπάρχουν και κάποιοι που απουσιάζουν και θα έρθουν μόνο σε αυτό το θέμα. Προτείνω να διακόψουμε μέχρι τις 11 όπως προβλέπετε. Uh, that's the planning, <laughs> ναι, αυτός είναι ο προγραμματισμός όμως. Οι άνθρωποι... Μάλιστα. Εντάξει, καλά τότε. Στις 11, ακριβώς όμως. Να είστε όλοι πίσω. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Είχαμε αυτή την σύντομη διακοπή, αλλά είμαστε έτοιμοι τώρα να συνεχίσουμε, γιατί είπαμε ότι στις 11 θα συνεχίζαμε τη συνεδρίασή μας, καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τον κύριο Χάστινγκς που είναι ο διευθυντής αυτής της αρχής της Εποπτείας Προστασίας Δεδομένων, ο Ευρωπαίος Επόπτης Δεδομένων και το βοηθό του κύριο Γιάννη Μπουταρέλη. Τους καλωσορίζουμε και περιμένουμε να μας παρουσιάσουν την ετήσια έκθεση του 2010 και μετά να τη συζητήσουμε χωρίς άλλη χρονοτριβή. Σας δίνω το λόγο κύριε Χάστινγκς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τις αδερές γραμμές της έκθεσης και τα κυριότερα σημεία της ε, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Έχετε λάβει ήδη σε αρχαίο PDF την έκθεση και περιμένουμε τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Η έκθεση δείχνει ότι το 2010 ήταν μια πολύ δυναμική παραγωγική χρονιά για την, εποπτεία, για την προστασία δεδομένων και για τον επόπτη. Πολύ δυναμική και φορτωμένη χρονιά. Κάτι που ευθυγραμμίζεται πλήρω και με την ανάγκη να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια πιο αποτελεσματική προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και των προστατικών δεδομένων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Γιατί υπάρχει όλο και μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση, κυριαρχία του διαδικτύου και εκτεταμένη χρήση του και παρέμβαση σε όλα τα στοιχεία της ζωής, ακόμη και στα πιο ιδιωτικά. Και αυτή η τάση μας αγγίζει όλους. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις δραστηριότητες της διοίκησης να εντείνει τις προσπάθειές της. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι δύο τρίτα όλων, του συνόλου των Ευρωπαίων πολιτών ανησυχούν ή ανησυχούν σοβαρά για την προστασία της ιδιωτικής του ζωής και των προσωπικών τους δεδομένων. Σε μερικές χώρες μάλιστα ο αριθμός αυτός είναι ακόμη πιο σημαντικός. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 92% του πληθυσμού με βάση την ετήσια έρευνα της ε, Βρετανικής ε, Υπηρεσίας Ενημέρωσης ανησυχεί για την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων. Βλέπετε τι ορολογία χρησιμοποιείται. Και μάλιστα ο αριθμός αυτός ε, αυξάνεται συνεχώς και η ανησυχία αυτή για την προσωπική ζωή και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται στη δεύτερη θέση των ανησυχιών των πολιτών πια. Το ίδιο και στην Γερμανία και στην Αυστρία. Γιατί λοιπόν ε, αυτή η τάση, αυτή η ανησυχία. Γιατί η όλο και μεγαλύτερη μας εξάρτηση από την πληροφορική και την επικοινωνία υπάρχει... οδήγησε ταυτόχρονα σε αύξηση των Τη ανάγκη για προστασία των δεδομένων. Έχουμε και τον αντίκτυπο τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Η συνθήκη τη Λισαβόνα έδωσε μια στέρη νομική βάση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής, ακόμη και αυτούς που δεν περιλάμβανόνται στον πρώην πρώτο πυλώνα. Γι' αυτό και η προστασία των δεδομένων είναι όλο και πιο σημαντικό θέμα και βρίσκεται στο επίκεντρο των ε, ενωσιακών πολιτικών. Και φυσικά εσείς, ε, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, το γνωρίζετε. Συνεχίζεται και η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Νομικού Πλαισίου για την Προστασία Δεδομένων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει την πρόταση για ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο και θα ψηφίσει, δεν κάνω λάθος, ε, αυτή τη βδομάδα την αρχική υποστήριξη και θα υποβάλλεται και προτάσεις για την αναθεώρηση αυτή. Η αναθεώρηση αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια φιλόδοξη πρόταση που θα ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες που δημιούργησε η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει η πρόταση αυτή να δίνει τη βάση για μια πιο αποτελεσματική προστασία προσωπικών δεδομένων σε μια στην μελλοντική κοινωνία της πληροφορίας. Ε, ε, για τα επόμενα χρόνια και μετά το 2020. Φυσικά ε, και το, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, ε, η, ατζέντα, η ψηφιακή ατζέντα αλλά και το πρόγραμμα για την βιώσιμη και συμμετοχική ανάπτυξη ασχολούνται με το θέμα αυτό. Και μάλιστα η ιδιωτική ζωή και η προστασία των δεδομένων βρίσκονται στο επίκεντρο και της παγκόσμιας προσοχής όσα, για παράδειγμα, πρόσφατα ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, το ίδιο και οι και το Μάιο στην τελική τους διακήρυξη οι G8 αναφέραν την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Αναφέρθηκε ε, αυτό σημαντικό, ε, σημαντικός τρόπος για να κερδίσει κανείς την εμπιστοσύνη των χρηστών. Έχουμε μια σημαντική ευκαιρία λοιπόν και πιο αποτελεσματική προστασία της, ε, των προσωπικών δεδομένων. Να χρησιμοποιήσουμε φυσικά και αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες για να δούμε τις δραστηριότητές μας για το 2010 σε ό,τι αφορά την εποπτεία. Πέραν μια σειρά πιο διεξοδικών δραστηριοτήτων, υιοθετήσαμε και μια, ένα σημαντικό έγγραφο πολιτική με τίτλο Την παρακολούθηση και την εξασφάλιση συμμόρφωση με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Η πολιτική αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού. Μέχρι πέρυσι περιοριζόμασταν στο να υποβάλουμε συστάσεις και να ενθαρρύνουμε τη συμμόρφωση. Δεν προειδοποιούσαμε, δεν επιπλήταμε ή δεν επιβάλαμε δεσμευτικές υποχρεώσεις. Μετά από μια πενταετή ισχύ του κανονισμού πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εθετήσουμε μια πιο αποφασιστική στάση σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση και να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη συμμόρφωση των αρχών της προστασίας δεδομένων. Νέα πολιτική περιλαμβάνει και διάφορα κριτήρια για μια ενεργή διαφανή και συνεπή εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού. Ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι και το πεδίο εφαρμογής της εποπτείας αυξάνεται. Μετά την θέση σε ισχύ της ηθίκης των δεδομένων, ο κανονισμός 45-2001 για την προστασία των δεδομένων ισχύει όχι μόνο για τα κοινοτικά θεσμικά όργανα ε, και για τις ενέργειές τους εντός του κοινοτικού δικαίου ισχύει πια σε όλα τα ευρωπαϊκά κοινοτικά θεσμικά όργανα και φορείς ακόμη και για τομείς που εκπίπτουν ε, των αρμοδιοτήτων του κοινοτικού δικαίου εκτός και αν φυσικά άλλες ε, ευρωπαϊκές διατάξεις ρητά, και το τονίζω αυτό, ρητά προβλέπουν κάτι διαφορετικό. Οι ακριβείς συνέπειες αυτών των αλλαγών για τις εποπτικές δραστηριότητες του επόπτη εξετάζονται και μάλιστα έχουμε συνεχίσει επαφές με τους αρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς. Υπάρχει και το δίκτυο των αξιωματούχων προστασίας δεδομένων που αυτή τη στιγμή καλύπτει 50 φορείς και σώματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το δίκτυο, εντυπωσιακό και τον Οκτώβριο το δίκτυο αυτό ε, αποκριστάλλωσε ένα πολύ σημαντικό έγγραφο σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες των αξιωματούχων προστασίας δεδομένων στα ευρωπαϊκά ε, και άλλα όργανα που εμπίπτουν στον κανονισμό. Και μάλιστα το γραφείο του επόπτη το ενέκρινε. Σε ό,τι αφορά τη διαβούλευση, συμμετέχουμε και σε διάφορες άλλες εργασίες για προσπάθεια εξυγχρονισμού του νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων. Σε πολλές περιπτώσεις ε, έχουμε προωθήσει φιλόδοξες προτάσεις για ένα σύγχρονο περιεκτικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων που θα καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και θα εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία των δεδομένων. Και μάλιστα ε, έχουμε εκπονήσει και δημοσιεύσει μια σχετική γνώμη τον Ιανουάριο με τις ε, λεπτομεριακές μας θέσεις. Ε, φαντάζομαι έχετε λάβει γνώση αυτού του εγγράφου το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και η ψηφιακή ατζέντα είναι άλλα σημαντικά προγράμματα με σημαντικές συνέπειες και για την προστασία των δεδομένων και θα τύχουν της δέουσας παρακολούθησης στα πλαίσια των, της διαβούλευσης. Η προστασία δεδομένων έχει αναδειχθεί σε βασικό στοιχείο νομιμοποίησης αλλά και αποτελεσματικότητας και για τους δύο τομείς. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι πέρυσι είχαμε αριθμό ρεκόρ 19 νομοθετικών πρωτοβουλειών για διάφορα θέματα, όπως την, την ατζέντα για την ευρωπαϊκή εσωτερική πολιτική, για την αντιδημοκρατική προσπάθεια, για τη μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, για διαχείριση πληροφοριών σε θέματα δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας, ε, ιδιωτική ζωή στο ψηφιακό πρόγραμμα και τη Συμφωνία Άκτα όλα αυτά τα θέματα θα απασχολήσουν και εσάς και όλες οι σχετικές γνωμοδοτήσεις υπάρχουν στο, στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Επόπτη. Και μάλιστα στην ιστοσελίδα μας έχουμε και ένα κατάλογο με τις διαβουλεύσεις που συμμετέχουμε και εκεί βρήκαμε 70, παραλαμβάνω 70 σημαντικά θέματα, εκ των οποίων 34 θεωρούνται ως προτεραιότητες. Έχουμε τρία χρώματα κόκκινο, κίτρινο και πράσινο, θα τα δείτε στην ιστοσελίδα. Θα αυτά τα 34 θέματα θα τα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγης και θα υποβάλουμε και σχετική γνωμοδότηση. Οπότε στο μέλλον θα αυξηθούν οι, τέτοιες, οι γνωμοδοτήσεις μας αυτές. Και ήδη έχουμε ξεπεράσει φέτος, τα μισά σχεδόν του έτους, το περσινό μας επίπεδο. Χαίρομαι για την προσοχή που δίνει η Επιτροπή, το Συμβούλιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ε, γνωμοδοτήσεις μας. Ακόμη και οι πιο επικριτικές μας γνωμοδοτήσεις ε, κρίνονται ως ευπρόσδεκτες ε, και επικοδομητικές από τα άλλα θεσμικά όργανα. Εν συντομία θα ήθελα να επισημάνω το ρόλο μας σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις. Για παράδειγμα, την αγωγή της, Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Γερμανίας 518-07. Εκεί το ΔΕΚ επισήμανε την ανάγκη απόλυτης ανεξαρτησίας της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων. Και μάλιστα αναφέρθηκε το, η σύσταση του γραφείου μας ως ε, βασική προδιαγραφή. Αναφέρθηκε όχι μόνο σε συγκεκριμένο άρθρο της Οδηγίας Προστασίας Δεδομένων Ομολογία, αλλά αναφέρθηκε και στο άρθρο 8 του, της Ευρωπαϊκής Χάρτας και το σχετικό άρθρο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομολογία αυτή του ΔΕΚ θα έχει σημαντική επίπτωση στο νέο νομικό πλαίσιο και ελπίζω ότι θα προσδιοριστεί περαιτέρω το νομικό αυτό πλαίσιο. Ανέφερα ότι στα πλαίσια της έκθεσης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που αν δεν κάνω λάθος σας υπευλήθη το πρωί, έγινε η σχετική παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης, έχουμε και το ρόλο των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων και ορισμένες αδυναμίες που επισημένονται καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για περισσότερη εναρμόνιση της θέσης των πόρων των εθνικών αρχών προκειμένου να έχουμε συνθήκες ε, ίσου ανταγωνισμού σε θέματα εποπτείας δεδομένων. Ανάγκη λοιπόν ε, στενότερης συνεργασίας και στα πλαίσια της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 Έχουμε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς και σε τέτοιες ομάδες επικεντρώσαμε την προσοχή μας στα θέματα στρατηγικής ε, σημασίας όπως την ερμηνεία βασικών διατάξεων της οδηγίας και την ε, συνεισφορά μας στην αναθεώρηση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου. Σημαντικό έργο έγινε και σε ό,τι αφορά το συντονισμό της ε, εποπτείας του συστήματος Eurodac. Εκεί ε, έχουμε κοινή αρμοδιότητα με τους εθνικούς φορείς. Το ίδιο μοντέλο ισχύει και για το σύστημα πληροφορίας για τα τελωνία. Και το ίδιο θα ισχύσει και ε, στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρίες και στο δεύτερο σύστημα ε, πληροφοριών Σέγγεν δεύτερης γενιάς, όταν τεθεί σε ισχύ. Και φυσικά όλα αυτά είναι χρήσιμα και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και ειδικά το θέμα της Eurodac. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον βοηθό μου, τον κύριο Τζοβάνι Μπουταρελή, να επισημάνει ορισμένες λεπτομέρειες και να σας εκθέσει τις βασικές μας προτεραιότητες για το μέλλον. Και κατόπιν, με μεγάλη χαρά, θα ακούσω τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας. Γενικά, αλλά και για την έκθεση πιο ειδικά. Ευχαριστούμε κύριε Χάστινγκ, ο κύριος Μπουταρελή. Ευχαριστώ αγαπητά μέλη. Η έκθεση του 2010 για το 2010 καλύπτει την έκτη συνεχόμενη χρονιά και τη δεύτερη χρονιά μέσα στα πλαίσια της τρέχουσας εντολής για την εποπτική αυτή αρχή. Όπως βλέπετε από τα 8 λεπτομερή κεφάλαια, εμείς ε, διαδραματίζουμε αυτό το ρόλο ως εγγυητή εγγυητής για την ένομη ε, κάλυψη και εξέταση δεδομένων. Άρα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει συστηματική εποπτεία των δικτών απόδοσης σε σχέση με όλους τους ε, ευρωπαϊκούς οργανισμούς με βάση το εγχείρημα που ξεκίνησε την άνοιξη του 2009 για την προστασία δεδομένων. Το έγγραφο ε, για την εποπτεία και τη συμμόρφωση ε, καλύπτει τις ε, διάφορες μορφές εποπτείας που ορίζει ο οργανισμός μας. Περιμένουμε λοιπόν, αναμένουμε από τους οργανισμούς να λογοδοτούν για οποιασδήποτε συστάσεις. Δηλαδή θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις ε, υποδείξεις και να μας το αποδείξουν. Εάν οποιοδήποτε δεν μπορέσει να δράσει, τότε θα πρέπει να προσφύγουμε με βάση τα ένδικα μέσα που διαθέτουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να δούμε ότι, μέχρι, ότι κατά, πόσο χρειάστηκε να προσφύγουμε σε κάτι τέτοιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να δούμε πού πρέπει να ανησυχούμε ε, για το ε, ρυθμό και βαθμό συμμόρφωσης των διαφόρων ιδρυμάτων και οργανισμών. Ε, αυτές οι εποπτικές και ε, καλύψεις έγιναν με βάση επιτόπιου, επιτόπιους ελέγχους. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι να ορίσουμε μία εποπτική αρχή. Το 2010 ορίσαμε 55 ελέγχους με ε, βάση εποπτεία με προειδοποίηση και 5 χωρίς ε, προειδοποίηση μέσα στο, στα πλαίσια του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και με βάση τις τυπικές αρχές για τις αξιολογήσεις και του προσωπικού. Συγκρίνοντας με το 2009 υπήρξε μία μείωση ως προς τους ελέγχους, τους συνολικούς ελέγχους. Γι' αυτό δεν έχουμε υπολοιπόμενες εργασίες, δεν έχουμε δηλαδή ε, εργασίες που, έχουν, ε, που από το παρελθόν και στις οποίες δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε. Έχουμε και 137 υποθέσεις που έληξαν διότι δώσαμε ε, συνέχεια στις προγενέστερες συστάσεις. Αναπτύσσουμε και άλλες μορφές εποπτείας όπου πως την διαχείριση των παραπώνων και των προσφυγών με βάση συγκεκριμένες θεματικές. Και βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η πολυπλοκότητα των υποθέσεων. Αν και έχουμε μείωση υποθέσεων κατά 15% είχαμε 94 υποθέσεις σε σχέση με ε, ε, πρόσβαση στα στοιχεία και απαλυφή στοιχείων. Τα δύο τρίτα αφορούσαν μη παραδεκτές και από τις 25 είχαμε μη συμμόρφωση, περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και υποβλήθηκαν και συστάσεις τους επόπτες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι διοικητικές ε, ε, εποπτείες και διαδικασίες παραπομπής σε πειθαρχικό, έτσι ώστε να βασιστούμε στην ε, βάση συμμόρφωση 45 2001. Επίσης, επιτελέστηκε περαιτέρω εργασία ως προς διοικητικά μέτρα και αποστήλαμε και μία επιστολή σε όλους τους αρχιεπόπτες και οργανισμούς για να ενημερώσουν τα στοιχεία τους, να τα επικαιροποιήσουν, υποστηρίζοντας την συμμόρφωση ως προς την προστασία δεδομένων, ως προς την ε, διαδικασία διαβούλευσης. Μιλήσαμε για 19 ε, συμμορφώσεις και συμβάσεις νομοθετικού περιεχομένου, λαμβάνοντας υπόψη την ε, ψηφιακή ατζέντα και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Η διεπαφή μεταξύ τεχνολογίας και ιδιωτικής σφαίρας ελήφθη υπόψη και αυτό που μας απασχόλησε είναι η ουδετερότητα του διαδικτύου και των δικτύων με βάση τον ε, ε, τις αποφάσεις This opinion adopted on uh, items which are every day in your agenda, the EU, US internet. Έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη το, την προστασία δεδομένων με την άκτα 2 ε, στοιχεία διάδοσης επιβατών και εφαρμογή των δεδομένων στην εσωτερική αγορά. Ήρθαμε σε επαφή με όλους τους συναδέλφους έτσι ώστε να ασχοληθούμε με βασικά στοιχεία προστασίας δεδομένων και συνεισφέραμε θετικά σε ζητήματα όπως ε, ε, του ελεγκτή και του επόπτη. Μέσα στα πλαίσια τη Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων το 2010 είχαμε αύξηση του προσωπικού μας, γι' αυτό ασχοληθήκαμε με τον προγραμματισμό εσωτερικές διαδικασίες και εφαρμογή του προϋπολογισμού είχαμε επανοργάνωση της Γενικής μας Γραμματείας έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων μας. Βλέπετε το νέο οργανόγραμμά μας στο διαδίκτυο. Επίσης έχουμε καλύτερη ε, επικοινωνιακή πολιτική και εισήχθησαν και τα γερμανικά ως τρίτη γλώσσα εργασίας επιπροσθέτως των αγγλικών και γαλλικών στην επικοινωνιακή μας πολιτική. Ως προς τις προτεραιότητές μας για το 2011, ε, η αναθεώρηση της οδηγίας είναι μία από τις προτεραιότητες. Η Επιτροπή έχει εκδώσει μία έκθεση αξιολόγησης και στην πρόσφατη έκθεσή μας θεωρήσαμε ότι η οδηγία δεν καλύπτει τα θεμελιώδη δικαιώματα ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της αναλογικότητας. Θα συνεχίσουμε να εποπτεύουμε με βάση τα στοιχεία opt-in, στοιχεία τεχνολογιών εχμής, δυνάμει της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 2020 και μέσα στα πλαίσια της ψηφιακής ατζέντας θα λάβουμε υπόψη και άλλες πρωτοβουλίες μέσα στο πλαίσιο των μεταφορών και ανταλλαγής πληροφόριου ως προς ε, τη διαδικασία γενικότερης ενσυνειδητότητας θα δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων και θα έχουμε γραφα κατευθυντηρίων γραμμών για ιδιαίτερα εργαστήρια και σεμινάρια. Επειδή ως προσελέγχους ex post δεν υπάρχουν εργασίες που να έχουν μείνει πίσω, θα προσπαθήσουμε να έχουμε νέες διαδικασίες επεξεργασίας έτσι ώστε να υπάρχει λογοδοσία και προστασία του ιδιωτικού βίου από πλευράς δημοσίων διοικήσεων και θα εποπτεύουμε την προστασία προσωπικών δεδομένων με βάση τους νέους οργανισμούς και ένα ε, νέο στοχοθετημένο εγχείρημα ε, προστασίας των δεδομένων. Νομίζουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή δεδομένων η οποία έχει θεσμοθετική παντού, σε όλες τις δραστηριότητες μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καθώς και την Επιτροπή σας, διότι μας συνέδραμε και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και το προσωπικό μας. Ευχαριστούμε κύριε Χάστινγκς, κύριε Χάστινγκς και Γκουταρέλη για την έκθεση αυτή, για το ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη. Τώρα θα έχουμε ερωτήσεις από τα μέλη. Ο κύριος Δίαφ Ντεμέρα έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χάστινγκς τα εξής δύο θέματα που έφτιαξε στη σελίδα 59 της έκθεσης το κεφάλαιο 362 γίνεται λόγο για τη χρηματοδότηση της ε, ε τρομοκρατίας μέσα στα πλαίσια του ε, SWIFT και ως προς τις δραστηριότητες της Europol, η οποία βασίζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου και θα συνταχθεί ένας νέος κανονισμός. Το Συμβούλιο μπορεί να λάβει αποφάσεις σε σχέση με την προστασία των δεδομένων. Ως προς ε, την κοινή εποπτική αρχή, ξέρετε ότι υπήρξε μεγάλο θέμα με την αρχή του επόπτη και την διαβίβαση δεδομένων. Κύριε Χάστινγκς, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις με βάση την απόφαση του Συμβουλίου. Υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων στα πλαίσια της Europol ή όταν θα πρέπει να συντάξουμε το νέο κανονισμό για τη Europol θα πρέπει να εισαγάγουμε ε, μηχανισμούς για να υπάρχει καλύτερη ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων. Η κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τους κυρίους Χάστινγκς και Μπουταρέλη για τη δραστηριότητά τους εδώ και αρκετό καιρό και για τη σημερινή παρουσίαση. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι εσείς μέσα στα πλαίσια της εποπτικής αρχής είσαστε, αποτελείτε ένα από τα προσφυλή μας θέματα στο Κοινοβούλιο αλλά και στην Επιτροπή αγάπη μας ιδιαίτερα, διότι αναφερόμαστε πάντα σε εσά όταν χρειαζόμαστε διασαφήσεις και όταν θέλουμε να γνωρίσουμε τι οδό, ποια οδό θα πρέπει να ακολουθήσουμε, όχι επειδή έχετε ε, μία ε, προσέγγιση καθαρά διαδικαστική, δηλαδή διευθέτησης διαφορών στην προσέγγισή σας, αλλά επειδή σας ενδιαφέρει πραγματικά η προστασία των δεδομένων. Δεν έχετε δηλαδή δικονομική προσέγγιση. Μιλήσατε για πολλά θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων σας. Καλύψατε ένα ευρύ πλαίσιο. Μιλήσατε για τη Frontex. Το ίδιο μας απασχολεί με στα πλαίσια της Eurodac και την θέσει σε ισχύ αυτό τον, μάλλον την εφαρμογή αυτών των δεδομένων. Το θέμα του PNR εκρεμεί τώρα στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα, δηλαδή ο αποκλεισμός του διαδικτύου και άλλα θέματα. Απλώς αναφέρομαι σε μερικά. Επειδή ορισμένες από αυτές τις οδηγίες και αναδιατυπώσεις καθώς και αναθεωρήσεις βασίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου, διότι από τη μία πλευρά βρισκόμαστε εμείς, από την άλλη όμως το Συμβούλιο. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα πείσετε το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη τα δικά σας δεδομένα τα δικά σας λεγόμενα. Πώς μπορείτε να τους πείσετε. Γιατί όλα αυτά τα θέματα που προανέφερα βρίσκονται επιτάπητος και μας απασχολούν ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας τον κύριο Χάστινγκς και τον κύριο Βουταρέλη για την παρουσίαση. Σίγουρα αξίζει ε, η προσπάθειά σας αναγνώριση όπως είπε και η κυρία Βέμπερ και σε πολλούς τομείς φαίνεται ε, η έκθεση απολύτως δικαιολογημένη. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση για ένα συγκεκριμένο σημείο. Γιατί ε, δεν συζητήσαμε ακριβώς για τα δεδομένα των επιβατών. Διαβάζω στην έκθεσή σας ότι ιδιαίτερα το θέμα της ανάλυσης κινδύνου και του λεγόμενου profiling ε, είναι, λέτε, προβληματικό. Και θα με ενδιέφερε πολύ να μάθω εκεί. Υπάρχουν ε, κάποιες προσπάθειες επίλυσης, ενασχόληση με αυτό το θέμα. Γιατί αυτό ισχύει και για τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εξ όσων βλέπω εδώ ε, και με την Αυστραλία. Και είναι ε, έτσι κομβικό σημείο, κεντρικό για τις ανάλυσεις σας. Κάποιες ε, συγκεκριμένες συμπεριφορές, καμιά φορά ταυτίζονται με συμπεριφορές υπόπτων. Και αυτό δεν είναι ε, μεμονωμένο, δεν είναι τυχαίο, βασίζεται σε πολλές πληροφορίες. Και σας ερωτώ, έχετε κάνει σκέψεις για το πώς ε, θα μπορέσετε να το ορίσετε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now, Mr. Voss. Ευχαριστώ κύριο Βος. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πολλά μικρά ερωτήματα. Πρώτον, Επεξεργαζόμαστε αυτό το καιρό την οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Και ένα σημείο βασικό είναι η ενιαία εφαρμογή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό το θέμα το επιγραμμικό ή μη επιγραμμικό online, offline είναι αρκετά καθόδες και για την προστασία δεδομένων. Και χρειάζονται σαφείς κανόνες. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Υπάρχει καμιά δυνατότητα παντού στην Ευρώπη να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο το δίκαιο για την προστασία των δεδομένων. Ή ε, υπάρχουν διαφορές πάγιες και μόνιμες. Αυτές οι διαφορές που βλέπουμε σήμερα είναι ε, προσωρινές ή όχι, γιατί θέλουμε στο μέλλον να εφαρμόζονται αυτά ενιαία. Ένα δεύτερο, στην ίδια μου τη χώρα, τη Γερμανία, στο μεταξύ έχω την εντύπωση ότι ε, το παρακάνουν στην προστασία των δεδομένων. Δηλαδή, στο μεταξύ, θέλουν λέει, να προστατεύουν και ανώνυμα δεδομένα, που δεν είναι καν προσωπικά αφού είναι ανώνυμα. Και δεν καταλαβαίνω. Αν μπούμε σε μια ρύθμιση που συγχαίει τα σύνορα και τα όρια, μήπως βοηθήσουμε και οδηγήσουμε σε συνολική σύγχυση στον πληθυσμό, ε, όταν το παρακάνουμε στις λεπτομέρειες να σας δώσω ένα υπερβολικό παράδειγμα, πραγματικά πάρα πολύ υπερβολικό. Ας πούμε να έχουμε διαφορετικές ε, μορφές προστασίας των δεδομένων για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες. Σας λέω ότι υπερβάλλω. Ε, γιατί νομίζω ότι το παρακάνουμε στη προστασία δεδομένων και χάνουμε το μέτρο. Στη συνέχεια, η προστασία των δεδομένων και ασφάλεια είναι κάτι που συζητούμε μαζί. Συνδεδεμένα και τα δύο δηλαδή αυτά πώς συνδέονται μεταξύ τους η σημερινή μας ψηφιακή πραγματικότητα. Καμιά φορά μπορεί να αυξηθεί και η ασφάλεια με τη χρήση κάποιων δεδομένων. Και από το πρόγραμμα TFTP που λέμε ότι διαβάζουμε υπερβολικό αριθμό στοιχεία. Μήπως θα πρέπει να έχουν οι Ευρωπαίοι ένα δικό τους πρόγραμμα ξεχωριστό για να απαντούν σε μεμονωμένα αιτήματα ή ερωτήματα και να διαβιβάζουν μόνο αυτό που τους ζητάνε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Νετσβάλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπαίνω κι εγώ στο χώρο εκείνων που ευχαρίστησαν ε, τον επόπτη προστασίας δεδομένων και μάλιστα με επένους και συμφωνώ γιατί πραγματικά κάνετε τη εργασία και ξέρετε έργο και την τελευταία επταετία έχετε στήσει έτσι αυτή την ε, ε, αρχή που είναι πολύ μεγάλο ατού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω μια μικρή ερώτηση, πολύ απλή. Συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνεται σε εσάς στη διαδικασία προετοιμασίας ε, νομοθετικών προτάσεων. Εσείς είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει υπόψη της ε, στην νομοθεσία Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις δικές σας συστάσεις. Γιατί έχω υπόψη μου μια συγκεκριμένη περίπτωση που είναι αξιολόγηση της οδηγίας για την ε, διατήρηση προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τη τόσο εξαιρετική εργασία πραγματικά και τη στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με την Επιτροπή μας. Από προσωπική εμπειρία πρέπει να πω ότι έχω φεληθεί πολύ ε, από τη συνεργασία ε, με το γραφείο σας στην ακαθόδη πραγματικά υπόθεση της Frontex που είχα φορτιστεί να επεξεργαστώ. πρώτη φορά έχουμε μια τέτοια μορφή αρχής επιβολής ε, του νόμου ας πούμε και προσωπικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η Frontex ασχολείται πάρα πολύ με προσωπικά δεδομένα. Μέχρι τώρα ε, πληρώνεται από Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες και μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να τα αξιοποιήσει αυτά τα στοιχεία γιατί ήταν θολό το τοπίο. Τώρα επιτέλους έχουμε μια διάταξη την οποία υποστήριξε ε, με ενθουσιασμό η Επιτροπή μας και θα πρέπει να συνεχιστεί. Ερωτώ λοιπόν, ο επόπτης προστασίας δεδομένων θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για άλλους οργανισμούς επιβολής του νόμου και μάλιστα για τη συνεργασία μεταξύ τους. Δηλαδή, τι εννοώ, θα πρέπει να έχουμε τέτοιους οργανισμούς επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να συνεργάζονται, να συνομιλούν, να μοιράζονται ε, πληροφορίε και εμπειρίες πάντα ε, στο στενό πλαίσιο του νόμου. Και μάλιστα με διευκρινήσεις που έχετε κάνει σε μεγάλο βαθμό εσείς οι ίδιοι. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Φλότρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, και εγώ θα προσθέσω τη φωνή μου ε, στους επένους και στις ευχαριστίες. Νομίζω ότι ε, θα φανεί υπερβολικό, αλλά είναι αλήθεια ότι οι γνωμοδοτήσεις σας θεωρούνται Ευαγγέλιο. Μπράβο σας. Λύνουν όλες τις διαμάχες και τους διαπληκτισμούς μεταξύ των πολιτικών ομάδων για τις τροπολογίες. Ακούμε με θρησκευτική ευλάβεια ε, τη γνώμη σας γιατί δείξατε με τον επαγγελματισμό σας άκρα αξιοπιστία και αυτό είναι πολύ αποφασιστικό για τη δουλειά μας. Επανέρχομαι στη Frontex, όπως είπε ο εισηγητής μας ο κύριος Μπουσουτήλ και εσείς συμβάλλατε πάρα πολύ στην επίλυση των προβλημάτων που είχαμε στις τροπολογίες και για να συμφωνήσουμε. Εγώ διαπίστωσα και ρωτάω αν μπορείτε να ψάξετε κάτι για τους ευρωπαίους οργανικούς οργανισμούς. Στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας και σε μια συνέντευξη του εκπροσώπου τύπου της Frontex διαπίστωσα ότι συλλέγουν στοιχεία από μόνοι τους ε, προσωπικά. Και το λένε και ανερυθρίαστα. Στα ελληνοτουρκικά σύνορα, χερσαία, υποδέχονται τους ε, μετανάστες και συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο με πληθώρα προσωπικών στοιχείων δεδομένων. Και το λέει πολύ ωραία σε μια βουλγαρική εφημερίδα ο εκπρόσωπος της Frontex που λέει στην Ιταλία έχουμε 10 με 15 ειδικού που ταυτοποιούν τους ε, μετανάστες και βοηθούμε τις Ιταλικές αρχές. Τι θα πει αυτό, αρκεί αυτή η ταυτοποίηση να γίνεται ε, για ε, προς όφελος ή κατόπιν αιτήματος ενός κρατικού οργανισμού και αυτό απαλλάσσει τη Frontex από την υποχρέωση να τηρεί την εντολή της και να μην κάνει τέτοια πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την αναθεώρηση της Frontex. Να δούμε ε, σε ποιο βαθμό αναλαμβάνουν ή δεν αναλαμβάνουν, αποποιούνται την ευθύνη τους. Από αυτή τη στιγμή εργάζονται για λογαριασμό κάποιες κρατικής αρχής ενός τρίτου κράτους. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάτφορτ. Ευχαριστώ. Δεν πρόκειται να παραλάβω αυτά που είπε η κυρία Φλότρ. Παρόλο που τα συμμερίζομαι, γιατί θα μετατραπούμε σε χορό εγκομείων εδώ πέρα, σε χώρο εγκομείων προ τον επόπτη. Πάντω, όλοι εκτιμούμε ιδιαίτερο το έργο του Ευρωπαίου Επόπτη προστασίας Δεδομένων. Έχω μία ερώτηση ως ό,τι αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών. Το γραφείο του Ευρωπαίου Υπόπτη θεωρεί ως τμήμα του ρόλου του τον εντοπισμό και την επισήμασης που μπορείτε να κάνετε στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, πιθανότητα αξιοποίηση υφιστάμενων πηγών δεδομένων αντί να συγκεντρώνουμε νέα δεδομένα, να αξιοποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό PNR, ασκείται πίεση για ένα εσωτερικό, ενδοκινοτικό PNR, για μια ενδοκινοτική συλλογή δεδομένων και μεταφορά στοιχείων επιβατών. Βέβαια, αν δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία ενδοκινοτικά PNR, ακούστηκε το επιχείρημα ότι θα υπάρχει από τους ελευθερεμπόρους, για παράδειγμα, ένα τρόπος παραμέρισμα θα, παρα, θα υπερκερνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όταν έρχονται από την Λατινική Αμερική στο Λονδίνο, για παράδειγμα, όταν ξέρουν ότι τους παρακολουθούν, θα πάνε μέσω Φραγκφούρτης και θα πάρουν μια εσωτερική πτήση. Σε τέτοια περίπτωση χρειάζεται συνεργασία μεταξύ της ε, γερμανικής αστυνομίας και των της υπηρεσίας συνόρων σε ό,τι αφορά την χρήση δεδομένων ε, από τρίτες χώρες, αντί να προβαίνουμε σε νέα συλλογή δεδομένων ενδοκινοτικά. Αυτό είναι ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα που θα μπορούσα να βρω. Και σε όλο το έργο που κάνατε για αναλογικότητα και αναγκαιότητα, Πιστεύετε ότι είναι σκόπιμο αντί να θεσπίζουμε νέα μέτρα με ενίσχυση της συνεργασίας να αξιοποιούμε τα υπάρχοντα. Και αν έχουμε καλύτερο συντονισμό και συνεργασία μπορούμε να χρησιμοποιούμε κοινά υπάρχοντα στοιχεία. Βέβαια υπάρχει το θέμα της πρόσβασης σε υπάρχοντα δεδομένα, αλλά θα χρειάζεται έτσι να προσφεύγουμε στην ε, συλλογή νέων δεδομένων, γιατί κάθε νέα συλλογή περιέχει και προβλήματα. Κυρία Ένστ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και από την πλευρά τη ΚΟΕ θα θέλαμε να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Χαστίν. Σε πολλά θέματα συνεργαστήκαμε. Κατά τα άλλα και σε θέματα που αφορούν το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπετε ερωτηματολόγιο των βοηθών και μας υποστηρίξατε, ακόμα και αν αποτύχαμε στην προσπάθειά μας αυτή. Αυτά εισαγωγικά. Θα ήθελα όμως να επανέλθω στα εξή τρία θέματα. Πρώτον, κανόνες για τον επόπτη και πλήρης ανεξαρτησία για τον επόπτη προστασίας δεδομένων. Το τονίσατε πάρα πολύ στα όσα μας είπατε και εύλογα. Υπάρχει και λόγος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν δεδομένη η ανεξαρτησία μπορείτε να μας πείτε έτσι πολύ συνοπτικά τι λείπει ακόμα και τι θεωρείτε πολύ σημαντικό από αυτά που λείπουν να εφαρμόζονται στην πράξη. Το δεύτερο, μας αφορά βεβαίως πάρα πολύ ε, όταν πρόκειται για τα χίδινη, τη, τη μαζική ε, αποστολή ε, στοιχείων. Μας αφορά και για το PNR και για το SWIFT, γιατί ο κίνδυνος του profiling είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το είπατε επανειλημμένα και στη δική σας έκθεση αυτό ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Πώς το αξιολογείτε αυτή τη μαζική αποστολή δεδομένων στο PNR και στο SWIFT. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε το στιγματισμό του profiling. Και το τρίτο αφορά την περίφημη προστασία των προσωπικών δεδομένων στους ερωτές σώματος. Πώς το βλέπετε αυτό και πώς θεωρείτε ε, ότι εξασφαλίζεται, αν εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων με τέτοια ε, μηχανήματα. Ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά για να ακούσουμε τις απαντήσεις των κυρίων Χάστινγκς και ε, Μπουταρέλη. Βέβαια, ακούσατε πολλές ερωτήσεις, ελπίζω. Να κάνετε μια προσπάθεια να τις συνοψίσετε γενικά στην απάντησή σας και να επικεντρωθείτε στα σημαντικότερα. Ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστώ θερμά για τις ε, ενθαρρυντικές σας παρατηρήσεις. Θα τις μεταβιβάσουμε φυσικά και στους συνεργάτες και το προσωπικό μας. Και φυσικά ευχαριστώ για τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας και αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε και θα τα αξιοποιήσουμε. Σε ό,τι αφορά τη σχέση με τη Europol, κύριε Ντίας Δεμέρα, η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει μια ειδική εποπτική αρχή που αφορά τα δεδομένα της αστυνομίας και μάλιστα αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ασχοληθούμε κυρίως με δεδομένα προσωπικού και να έχουμε στενή συνεργασία. Με αυτό ασχολείται τώρα το γραφείο μας. Βέβαια, το θέμα του συστήματος οικονομικού εντοπισμού τρομοκρατών εμπίπτει στο θέμα της ιδιωτικής ζωής και ρωτήσατε αν είναι ικανοποιητικά τα πλαίσια της προστασίας δεδομένων και οι ρυθμίσεις για τη Europol. Υπάρχουν αδυναμίες παντού. Η απόφαση για τη Europol υιοθετήθηκε πριν θέσει εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας, οπότε αναμένεται αναθεώρηση. Και στα πλαίσια της αναθεώρησης θα διορθώσουμε κάποια κενά και αδυναμίες και το πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προφανώς δεν επαρκεί και θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα της συνολικής αναθεώρησης. Κυρία Βέμπερ, λέτε ποια θα είναι η ακολουθητή στρατηγική για να πείσουμε το Συμβούλιο. Θα ξεκινήσουμε με μία σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση, τονίζοντας την ανάγκη ε, αποδείξεων με βάση την αναλογικότητα, την νομιμότητα, την επάρκεια των ερευνών και φυσικά τι εναλλακτικέ ε, λύσεις υπάρχουν. Αυτό στα πλαίσια της συζήτηση, όχι μόνο για την προστασία των δεδομένων αλλά και γενικότερα. Έχουμε συστηματικέ και τακτικέ επαφέ με τι διάφορε. και τις μελλοντικέ προεδρίες. Τώρα ήδη ξεκινήσαμε συναντήσεις με την Πολωνική Προεδρία και ιδιαίτερη Πολωνική Προεδρία ενδιαφέρεται για την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαίου από την προστασία δεδομένων σε διάφορα θέματα όπως είναι το PNR, προστασία δεδομένων και στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς κρατάμε βέβαια μια απόσταση αλλά βοηθάμε την κάθε Προεδρία με τα σχόλιά μας, την κριτική μας και την πρόταση εναλλακτικών λύσεων. Εγώ δεν είμαι απεσιόδοξος. Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής ίσως, αλλά νομίζω ότι η κατεύθυνσή μας είναι σωστή ακόμη και για το PNR. Και αυτό ρώτησε και ο κύριος Άλμπρεχτ. Και το profiling κινδύνου. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο σημείο ίσως. Αλλά γι' αυτό ακριβώ το λόγο προτείνεται και το καθεστώς PNR. Αν δεν υπάρχει σαφήνεια, αυτό είναι πρόβλημα της πρότασης. Θα πρέπει να υπάρχει τρόπος καταμέτρησης της αναλογικότητας, της παροχής εχεγγύων. Αυτά όλα θα πρέπει να τονιστούν. Το risk profiling μπορεί να είναι από κάποια άποψη προβληματικό και τα ιατρικά δεδομένα. Οι γιατροί κάνουν τέτοια ταξινόμηση των ασθενών για να δουν ποιοι χρειάζονται περισσότερης προσοχής, αλλά στην περίπτωση δεδομένων ο κίνδυνος να υπάρχει τέτοιο profiling κινδύνου και ταξινόμηση βάσει τον κίνδυνο είναι αρκετά προβληματικός. Και τι θα πει ακριβώς risk profiling. Επιλέχθηκε αυτός ο όρος για να ακούγεται πιο θετικά, αλλά νομίζω ότι προσπαθούμε απλώς να αποφύγουμε κάτι που όλοι ξέρουμε τι είναι. Αυτό που επιζητούμε είναι εχέγγυα, ώστε και οι αρμόδιες αρχές και ο επιβάτης να μπορούν να έχουν αντεπιχειρήματα. Γι' αυτό και θα πρέπει να επενδύσουμε σε μηχανισμούς που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, ούτε φυσικά έχουν διευκρινιστεί στην πρόταση. Γι' αυτό και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Κύριε Βός, θέσατε πολλές ερωτήσεις. Για παράδειγμα, πώς θα εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ομοιομορφία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ομοιομορφία και αρμονία μέσα στη διαφορά, στη διαφορετικότητα, στην ποικιλομορφία. Δεν θέλουμε να εξουδετερώσουμε οποιαδήποτε ποικιλομορφία. Αυτό θα ήταν και ασεβές. Αλλά απλώς θέλουμε να έχουμε περιορισμό αυτής της πυκλομορφίας που υπάρχει μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε πολύ διαφορετικούς τρόπους προστασίας δεδομένων, να εξασφαλίσουμε μια κάποια ομοιομορφία. Και αυτή είναι η ουσία της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα κοινό έδαφος για να προχωρήσουμε, όπως φάνηκε και από τη δική σας παρατήρηση. Οπότε το ζήτημα που ανακύπτει είναι σε ποιους τομείς χρειαζόμαστε ή θα προτείνουμε με περισσότερη ομοιομορφία ή περισσότερη ποικιλομορφία. Γιατί όταν έχουμε ποικιλομορφία και διαφορές, έχουμε περισσότερες ε, περιπλοκές και στην εφαρμογή του νόμου και στην επιβολή του νόμου. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Αυτή η πολυμορφία στην περίπτωση αυτή δυσκολεύει. Αν έχει υπερ, υπερεκτιμηθεί η προστασία των δεδομένων, μερικές φορές ναι. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ρεαλισμό πάνω απ' όλα γιατί δεν αρκεί να κάνουμε μεγαλεπίβολα σχόλια για την προσοχή των δεδομένων, πρέπει να την εφαρμόζουμε και εμπράκτος. Είναι υπερβολική ανάγκη προστασίας και ανώνυμων δεδομένων, όχι κατά ανάγκη. Το ίδιο και όταν συζητούμε για το risk profiling. Ίσως σε ορισμένε περιπτώσεις, ακόμη και για τα ανώνυμα δεδομένα, χρειαζόμαστε κάποιου μηχανισμού που θα στηριχθούν σε συστήματα αναλύσεων όχι βέβαια για μια συλλήβδη προστασία όλων των ανώνυμων δεδομένων, αλλά θα πρέπει και εκεί να προσδιορίσουμε πού βρίσκεται η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της ανάγκης προστασίας δεδομένων και της ανωνυμίας. Μέχρι στιγμής είναι καλή διαχωριστική γραμμή, ούτε υποβαθμίζουμε ούτε υπερτιμούμε την κατάσταση. Τώρα, ασφάλεια στην ιδιωτική ζωή. Το χρειαζόμαστε και τα δύο. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τέτοιους μηχανισμούς γιατί αν έχουμε ασφάλεια και πολύ ακριβή, ε, ε μάλλον ασφάλεις βάρος της ε, ιδιωτικής ζωής, ούτε και αυτό είναι καλό. Το πρόβλημα με το TFTP, το σύστημα οικονομικού εντοπισμού τρομοκρατών, είναι ότι η ασφάλεια της ιδιωτικής ζωής δεν ε, περιλαμβάνεται στα βασικά στοιχεία. Δεν ξέρω αν χρειάζονται αναθεωρήσεις του συστήματος αυτού του TFTP, Πάντως το ισχύον δεν είναι και πολύ ικανοποιητικό. Και αν το όντως θα προκριθεί ως τμήμα της λύσης το TFTP, το Σύστημα Οικονομικού Εντοπισμού του θα το εξετάσουμε. Κυρία Ινφέλτ, άτυπες διαβουλεύσεις. Γενικώ είμαστε ικανοποιημένοι από το πώς ε, λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις μας. Σε ό,τι αφορά την ε, παρακράτηση δεδομένων ή τη φύλαξη δεδομένων, εμείς ήμασταν πολύ επικριτικοί και ενθαρρύναμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε μια ισορροπημένη αξιολόγηση, κάτι που έγινε και θα είμαστε πολύ απαιτητικοί μέχρι ότου προταθούν σωστές λύσεις. Χαίρομαι για την ε, θετική αξιολόγηση της εμπειρίας ε, του κ. Μπουσουτήλα από τη Frontex. Και φυσικά δεν θα πρέπει να γίνεται ένα απλό copy-paste, και επικόλυση, αλλά η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αστυνομικών αρχών, γιατί όχι. Πολύ θετικά ήταν τα σχόλια και της κυρίας Φλότρ. Κυρία Λάτφορτ, για τη διαχείριση των πληροφοριών ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου Επόπτη. Είχαμε συνεργασία με τη Σουηδική Προεδρία και έκτοτε προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε μία μεθοδολογία όπου παρακολουθούμε τον τρόπο εφαρμογής και υποβάλλουμε και λεπτομερικές ερωτήσεις για το αν εξετάστηκαν δεόντως οι εναλλακτικέ λύσεις και ενδεχομένω μπορεί και εμείς να προτείνουμε ορισμένες τέτοιες εναλλακτικέ λύσεις. Δεν θέλουμε όμω εμεί συστηματικά να προβάλλουμε εναλλακτικέ λύσεις. Απλώς θέλουμε να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιστική στα επιχειρήματα και να επιμείνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν δεν έχουν εξεταστεί όλες οι εναλλακτικέ. Και κυρία Ένστ, η ανεξαρτησία είναι κέρια σημασία και το τονίζει η κοινομολογία του ΔΕΚ γιατί η αρχή προστασίας δεδομένων θα πρέπει να είναι σε θέση να προβεί σε μία έντιμη ε, και δίκαιη αξιολόγηση. Δεν θα πρέπει να επεμβαίνει κανένα στο έργο της προκειμένου να βρει τη σωστή ισορροπία η κάθε εποπτική αρχή και θα πρέπει να υπάρχει ισοτιμία μεταξύ των ε, εποπτικών αρχών. Αλλιώς πώς δεν νοείται ο συντονισμός ή η συνεργασία. Για, αυτό ισχύει για το PNR για τους αρωτές σώματος. Εκεί όλοι ε, αναχαιτήσαμε σε προκαταρκτική φάση την ε, λήψη απόφασης. Τώρα βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί η τεχνολογία και σε μεγάλο βαθμό είδαμε ότι έχουν ληφθεί υπόψη κάποιες λύσεις που απορρέουν από την τεχνολογία και τελικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το εργαλείο κατάλληλα και νομίζω ότι έχει βελτιωθεί η, σχέση, η θέση μας. Τώρα, η γενίκευση της χρήσης αρωτών σώματος δεν θα ήταν χρήσιμο. Με τη χρήση των σαρωτών σώματος, ακόμη και στην διευρυμένη εκδοχή και πάλι έχουμε θέματα ε, διαχείρισης δεδομένων, οπότε θα πρέπει να ισχύουν οι ασφαλιστικές δικλίδες. Μόνο έτσι θα υιοθετήσουμε ισορροπημένες λύσεις. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που μου επιτρέψετε να ξεπεράσω και το χρόνο. Ευχαριστούμε κυρία Χάστινς που μας βοηθήσατε και συνοψίσατε τις απαντήσεις σας ομαδοποιώντας τις. Ο κύριος Μπουταρέλη για να συμπληρώσει κάτι αν θέλει, ναι. Στο ένα λεπτό που μου διατίθεται θα ήθελα να πω στην κυρία Βέμπερ ότι λάβαμε ένα ενθαρρυντικό γράμμα από το Συμβούλιο για να έχουμε πιο σταθερές σχέσεις ως προς τη συζήτηση των θεμάτων μας, όχι μόνο ακροάσεις, αλλά τακτές συναντήσεις και επαφές. Αν και δεν είμαστε μόνιμα μέλη των ομάδων εργασίας και δεν μπορούμε να παρευρεθούμε στις συναντήσεις της ΚΟΡΕΠΕΡ ή του Συμβουλίου. Η Προεδρία τόνισε την ανάγκη να, είναι, να είμαστε σε μεγαλύτερη και περισσότερη επαφή για τη συνέχεια στα θέματα αυτά. Ως προς το PNR θα ήθελα να πω ε, ότι το θέμα profiling ε, σχετίζεται το θέμα είπα PNR ε, αφορά μια πολιτική, γενικότερη πολιτική, έτσι ώστε να γίνεται ε, μια συνεχιζόμενη συζήτηση. Αυτό απαντώντας στον κύριο Άλμπρεχτ και θα ήθελα να πω ότι θέλουμε μεγαλύτερη υποστήριξη από εσάς που πιστεύω ότι θα την έχουμε. Εκτιμώ το μήνυμα της κυρίας Λάντφορτ. Δηλαδή δεν μιλάμε για δημιουργία νέας πλατφόρμας, νέων συστημάτων. Αυτό όμως θα ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος των συστημάτων μας και αυτό το έχουμε υπογραμμίσει σε πολλές ε, πρόσφατες γνωμοδοτήσεις μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε κύριοι Hastings και Μπουταρέλη για τα στοιχεία που μας δώσατε ως υπεύθυνοι του Ευρωπαίου Πόπτη Προστασίας Δεδομένων. Σας ε, αποχαιρετούμε και στη συνέχεια έχουμε την έκθεση Ρωμέβα για την ίση μεταχείριση. Πρόκειται για το σημείο υπαριθμών 8 και αφορά την ίση μεταχείριση προσώπων ανεξαρτήτως ε, θρησκείας, πεπιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Θα ακούσουμε την παρουσίαση του θέματος από τον κύριο Ραούλ Ρομέβα σε σχέση με την γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου που ε, εγκρίθηκε στις 2 Απριλίου 2009 κατά, την, ε, κατά τις εργασίες της Ολομελίας υπό την προηγούμενη νομοθετική θητεία με βάση τη διαδικασία διαβούλευσης. Όμως η θέση εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας οδήγησε σε μια αλλαγή διαδικασίας σε σχέση με αυτό το θέμα με βάση τη διαδικασία συνένεσης και με βάση το άρθρο 9 της συνθήκης. Ο κύριος Ρωμέβα είναι ο εισηγητής αυτής της διαδικασίας συνένεσης της σύμφωνης γνώμης και η ε, Ουγγρική Προεδρία αποφάνθηκε επίσης επί του θέματος. Ελπίζω η Επιτροπή επίσης να παρουσιάσει τη θέση της με βάση εξελίξεις και οι βουλευτές μπορούν να λάβουν το λόγο για να παρέμβουν επί του θέματος. Θα ακούσουμε από τον εισηγητή, μετά το Συμβούλιο και μετά την Επιτροπή. Ρωμέβα. Ευχαριστώ. Δεν έχω τίποτα το ιδιαίτερο να προσθέσω ως προς τη συζήτηση αυτή. Πρόκειται για ένα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει εδώ και πολύ καιρό και έχει αποκλειστεί σε επίπεδο συμβουλίου, διότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν θέλουν να προβούν σε αλλαγές. Εάν όμως μελετήσουμε προσεκτικά το περιεχόμενο της πρότασης και τον κατεπήγοντα χαρακτήρα αυτής της πρότασης, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι κατανοητό γιατί δεν έχουμε μία συγκεκριμένη πρόταση επιτάπητος για να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο. Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν είχαν γίνει διαβουλεύσεις, αλλά χωρίς να μπορέσει να παρέμβει το Κοινοβούλιο νομοθετικά. Τώρα όμως ε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο διότι με βάση τη διαδικασία συμφωνής γνώμης μπορούμε να αποφανθούμε. Ε, ο κύριος And working, uh, quite closely. Η κυρία Μπέτεμβεχ είχε μπορέσει να αποφανθεί στα πλαίσια της προγενέστερης της προηγούμενης θητείας, αλλά μετά την Βελική Προεδρία παρενέβησαν και άλλες προεδρίες που δεν ήταν και τόσο ανοιχτές προς νέες προτάσεις, τις οποίες ε, δεν θεωρούσαν τόσο πρόσδεκτες σε σχέση με την τακτική συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Υπάρχουν τρία ερωτήματα λοιπόν προς το Συμβούλιο επί του θέματος και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο υπάρχουν απαντήσεις, διότι από όσο καταλαβαίνω υπάρχουν θέματα τα οποία σχετίζονται με το θέμα μας. Ακούσαμε σήμερα το πρωί τον υπεύθυνο της Οργάνωσης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη ανάγκη για την σύνταξη μιας οδηγίας προς αυτή την κατεύθυνση η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο πίεσης από τα κράτη-μέλη για να πείσουν τα άλλα ε, κράτη-μέλη έτσι ώστε να αρθεί αυτός ο αποκλεισμός σε επίπεδο Συμβουλίου. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω το Συμβούλιο πώς αντιλαμβάνονται αυτή τη γνωμοδότηση. Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τη νομική διάσταση του ζητήματος με ε, βάση την ε, κύρωση της ε, Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με πρόσωπα με αναπηρίες στην αρχή της Ουγγρικής Προεδρίας. Θα ήθελα να πω γιατί υπάρχει αυτή η επιφύλαξη από κράτη-μέλη, έτσι ώστε να κυρωθεί στην πράξη και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό αποτελεί μεγάλη αντίφαση και θα θέλαμε να απασχολήσει το Συμβούλιο με σαφήνεια. Επίσης, στο Συμβούλιο, στην Ομάδα Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων, υπάρχει μία ε, παλινοδία σε σχέση με το κεκτημένο ως προς άτομα με αναπηρίες, γιατί ε, αναφέρθηκε Αναφερθήκαν στο γεγονός ότι αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να ισχύσει για εργαζόμενους με ε, σύμβαση ας πούμε ορισμένου χρόνου αυτό το θέμα θα συζητηθεί και στο ε, Κοινοβούλιο. Όπως αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απίφθηνα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια είναι η θέση της επί του θέματος. Αυτά επί του παρόντος είμαι σίγουρος ότι και άλλοι συνάδελφοι θα υποβάλουν συμπληρωματικές ερωτήσεις και θέλω να ακούσω τι θα μας πούν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση του θέματος την παρούσα στιγμή. Θα ακούσουμε και την Κομισιόν και το Συμβούλιο και την Ουγγρική Προεδρία. Υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλο ένα θέμα που θα μας απασχολεί σήμερα το πρωί σε σχέση με μια συνάντηση, τη συνάντησή μας ε, in camera και κλεισμένο των θυρών. Και ελπίζω να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια από πλευράς ε, χρόνου, γιατί έχουμε και ένα μακρύ κατάλογο μελών. Θα κλείσουμε και τον κατάλογο αφού ακούσουμε από την Προεδρία ο κύριος Άντρας Λάσλο ή ο κύριος Ατίλα Φούλοπ. Κάποιος από τους δύο μπορεί να λάβει το λόγο εξ ονόματος της Ουγγρικής Προεδρίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εξ ονόματος της Προεδρίας. Με χαρά ήρθαμε να σας ενημερώσουμε για την οδηγία ε, κατά των διακρίσεων ή την οδηγία για την ίση μεταχείριση προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας, πεπιθήσεων, απειρίας, ηλικίας, γενετησίου προσανατολισμού. Για να σας ενημερώσουμε τι έχει γίνει στο Συμβούλιο. Όπως ακούσαμε ήδη, από το 2008 και συγκεκριμένα τον Ιούλιο, το 2008 έχει κατατεθεί αυτή η οδηγία. Τρία χρόνια μας απασχολεί και από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας χρειάζεται ομόφωνη απόφαση για να τεθεί σε ισχύ η οδηγία αυτή. Ξέρετε ότι το φάσμα είναι ευρύτατο και η προοπτική σε αυτό το θέμα. Και το θέμα εδώ δεν είναι η απασχόληση, αλλά η κοινωνική ασφάλιση ε, και άλλα θέματα στέγασης, παιδείας και πολλά ακόμα. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα λίγο να πω στην προϊστορία. Η Βελγική Προεδρία το Νοέμβριο του 2010 αξιολόγησε τη δράση της και την εργασία της και προσπάθησε ε, η Ουγγρική Προεδρία να ολοκληρώσει το θέμα, όπως μας είχε διαβιβάσει η προηγούμενη Προεδρία. Γνωρίζαμε από την αρχή ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το ζήτημα αυτό, γιατί διότι υπάρχουν κίνδυνοι. Αντιδρούν τα κρατη για λόγους ε, επικουρικότητας, αναλογικότητας ή ακόμα και αβεβαιότητας. Ε, όταν προσπαθούσαμε να εκπονήσουμε αυτή την οδηγία και να την προωθήσουμε. Η Βελγική Προεδρία ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα οικονομικά και τα θέματα της στέγης και εμείς επικεντρωθήκαμε σε άλλα πλέον. Πάντα με βάση αντικειμενικά στοιχεία ε, και επικεντρωθήκαμε ε, σε θέματα ατόμων με αναπηρία. Γιατί ιδιαίτερα σε αυτά τα θέματα, διότι αφορούν πάρα πολύ κόσμο, 70 με 80 εκατομμύρια, που είναι 10 με 15% του ε, κοινοτικού πληθυσμού. Επιπλέον, οι διατάξεις οδηγίας αυτής έχουν ως στόχο βεβαίως πάντα τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των προσώπων αυτών. Αυτή η ομάδα στόχος δηλαδή μπορεί να φτάσει σε καλύτερα βιωτικά επίπεδα και περισσότερη ευημερία. Αυτοί οι στόχοι πρέπει να σας πω εγγράφονται και στη στρατηγική 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είναι ο στόχος. Το 75% των ατόμων με αναπηρία να βρίσκουν καλύτερη απασχόληση, γιατί σήμερα είναι σε πάρα πολύ άσχημη μοίρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια στρατηγική μεγαλύτερη συμπερίληψη και ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Ε, φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να μπω στα εξής δύο σημαντικά για μένα θέματα. Πρώτον, προσαρμογή των ατόμων με αναπηρία και επίσης κατανομή του βάρους. Δεν μην πω σε λεπτομέρειες τώρα για την ουσία των θεμάτων αυτών, αλλά κατά τη διάρκεια των εργασιών μας ασχοληθήκαμε θέματα όπως το πώς μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο ή στην εθνική ενόμη τάξη της κάθε χώρας αυτή η προσαρμογή της κοινωνίας Έχει νόημα συστηματικής καταγραφής ε, των ε, διαφόρων ε, προβλημάτων και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση γενικά. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βοήθειά της. Χρειάζεται υποστήριξη αυτή η προσπάθεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε και για τις βασικές έννοιες, για τον ορισμό, Αλλιώ δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Τώρα, σε αυτά τα λίγα λεπτά που έχουμε δεν μπορούμε να πούμε ε, όλες τις λεπτομέρειες. πρέπει να σας πω ότι σε πολλά συστήματα στην ένωμη τάξη δηλαδή των κρατών μελών υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αλλά αυτή η ε, λογική προσαρμογή των συστημάτων επί της αρχής είναι κοινή ε, ομολογία αλλά αυτά που ισχύουν σήμερα ε, διαφέρουν πάρα πολύ από χώρα σε χώρα και σε ό,τι αφορά την παιδεία ή τη δημόσια διοίκηση κτλ. Η αρχή αυτή της λογικής ε, προσαρμογής ε, είναι κάτι που βλαβάνεται και σε ένα ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Ε, στόχος μας ήτανε η προσαρμογή αυτή να γίνει σταδιακά και να υπάρχει παντού δεδομένη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Δηλαδή, υπάρχουν από τη μια υποχρεώσεις που πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη όταν παίρνουμε αποφάσεις. Να συμφωνήσουμε για το πώς έχουν οι ορισμοί ε, και να εξηγούμε τι είναι αυτά με συγκεκριμένα παραδείγματα να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το πράγμα της λογικής προσαρμογής. Έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα, γιατί είναι αρκετά ασαφές. Και να σας μιλήσω και για τη δυσανάλογη κατανομή του βάρους. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα πρόσωπα με αναπηρία, αλλά ε, με ολόκληρη την οικονομία και μάλιστα την κάθετη διάταξη της οικονομίας. Εξετάζεται η οικονομική τους κατάσταση, οι δυνατότητες, ε, τα προσόντα, οι δεξιότητες, το δυναμικό που εμφανίζουν. Ελπίζω ε, με τον τρόπο αυτό να διευκρινίσαμε πολλά θέματα. Ε, κάναμε πρόοδους και προσβλέπω και στη μελλοντική συνεργασία μαζί σας. Και να, να συνεχιστεί η προσπάθεια στην επόμενη Προεδρία. και η Πολωνική Προεδρία είμαι βέβαιο θα ε, ασχοληθεί με αυτό το θέμα και αυτό που έχει σημασία είναι το πεδίο εφαρμογή νέα είναι έτσι ορισμένο ώστε να μην δίνει βάση για παρεξηγήσεις και να καταλάβουμε ότι οι υποχρεώσεις ισχύουν προ όλου. και αφορούν όλους. Και θα πρέπει να τα λέει αυτά ρητά η οδηγία. Τέλος, να ευχηθώ Καλή επιτυχία στην Πολωνική Προεδρία, στην εκπόνηση της οδηγίας αυτής. Και ευχαριστώ όλους όσοι παρακολούθησαν το θέμα αυτό μέχρι σήμερα και ελπίζω να συνεχιστούν και στην επόμενη Προεδρία η διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Φερνάντο Περέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά προτείνω να θυμίσουμε ότι πρέπει να συνοψίζουμε. Κανονικά η κυρία Λεμπάγε πρέπει να περιμένει απ' έξω για να μας κάνει την παρουσίασή της και έχουμε καθυστερήσει η Επιτροπή. Euh, Ευχαριστώ. Δεν ε, θέλω να περιμένει για πολλή ώρα η Γενική Διευθύντρια. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικό. Ευχαριστώ την, Ογγρική την Προεδρία για το έργο τελευταίο τελευταίου εξαμήνου. Όπως είπε ο κύριος Υπουργός, προσπαθήσαμε να βρούμε κάποια μέτρα για τις ε, απαραίτητες, ε, λογικές μάλλον, ε, διαρρυθμίσεις για τα άτομα με αναπηρία. Και αυτό είναι βασικό στοιχείο της οδηγίας. Οποιαδήποτε πρόοδος στο θέμα αυτό είναι πολύ σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρθηκε, στήριξε τις προσπάθειες της Ουγγρικής Προεδρίας και πιστεύουμε, όπως πολλές αντιπροσωπείς στο Συμβούλιο, ότι οι προτάσεις που έγιναν μετά την εξάμηνη συζήτηση είναι θετικές. Για να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Ρωμέβα για τις ε, μακροχρόνιες ενοχικές σχέσεις, εμείς δεν μπορούμε να περιορίσουμε τη, την εμβέλεια αυτού αυτής της πρότασης για τη λογική διαρρύθμιση, τις λογικές διαρρύθμισεις που πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι δεν είναι μυστικό ότι ε, το Συμβούλιο ακόμη πόρα απέχει από την ε, ε, απόφαση και η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν επηρεάζει την κατάσταση του Συμβούλου για το οποίο απαιτείται ομοφωνία. Αναφέρθηκε και ο ρόλος του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που πιστεύει ότι η οδηγία αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για να συμπληρωθεί το νομικό πλαίσιο πάταξης των διακρίσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, μας απογοητεύει αυτή η κολυσιεργία και η βραδύτητα με την οποία σημειώνεται πρόοδος. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την ανέβρεση τεχνικών λύσεων και μάλιστα θα ρίνουμε την επερχόμενη Προεδρία την Πολωνική να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει επαφές και γνωρίζουμε ότι η Πολωνική Προεδρία θα συνεχίσει την βάθηση σε τεχνικά ζητήματα των διατάξεων ΑΝΤΕΑΣ που επίσης είναι από τα επίμαχα σημεία της οδηγίας. Και φυσικά μπορεί και η Πολωνική Προεδρία να υπολογίζει στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανέβρεση τεχνικών λύσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί το ύψο επίπεδο νομικής ασφάλειας. Ασφάλειας δικαίου. Με την θέση ισχύ της συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να ε, εγκρίνει τη συμβαστική λύση του Συμβουλίου, να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του και από αυτήν την άποψη είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι συζητήσεις Συμβουλίου Κοινοβουλίου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και χαιρόμαστε που συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Καλώς θα ήθελα παρακαλώ οι ομιλητές να περιοριστούν στο 1,5 λεπτό γιατί ήδη έχει καταθέσει η κυρία Λεμπάη και δεν είναι σωστό να περιμένει, ούτε και μπορούμε να αναβάλουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Ο κύριος Κάσμαν πρώτα. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Η Ουγγρική Προεδρία μας είπε ότι υπάρχει πρόοδος και σαφήνεια. Εγώ δεν έχω τέτοια εντύπωση. Ούτε πρόοδος υπάρχει, ούτε και ενάργεια. Νομίζω ότι είναι τελείως σφαλμένη η αντίληψη του Συμβουλίου και δεν έχει καμία σχέση με την απασχόληση που καλύπτεται στην οδηγία πλαίσιο για την απασχόληση. Αν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα, κοιτάξουμε τι εθνικέ νομοθεσίε. Κοιτάξτε την νομοθεσία Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανία που έχουν ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Έλλειψη πολιτική βούληση παρατηρούμε, έλλειψη οράματο και έλλειψη θάρρου για τη διόρθωση τη κατάσταση. Και είναι τελείω εσφαλμένο αυτό το μήνυμα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελάχιστη δράση έχει αναλυφθεί σχετικά. Αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Αναπηρίες. Θα υπογράψουμε ε, και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εντός ολίγου. Και ουσιαστικά παραβιάζουμε αυτή τη συνθήκη και ε, είμαστε αντίθετοι και με την ε, σχετική νομολογία για την καταπολέμηση των διακρίσεων πρέπει να ανασκουμποθούμε και να λύσουμε τα προβλήματα. Λύθηκαν κάποια προβλήματα στην οδηγία ΡΕΙΣ. Αν υπάρχει πολιτική βούληση θα πρέπει να δούμε τι έγινε με την οδηγία για τις φυλές και τις εθνικότητες για σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες. Ήδη η οδηγία ΡΕΙΣ μας, δίνει, μας δείχνει το σωστό δρόμο. Και κάτι που λέω σπανίως. Ευτυχώς όμως που υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συνεχίζει να προωθεί και να προαγάγει τα συμφέροντα ανθρώπων που γίνονται θύματα διακριτικής μεταχείρισης άνευ λόγου και αιτίας και χωρίς καμία νομική θεμελίωση. Γιατί από το Συμβούλιο και τις Προεδρίες δεν έχουμε δει ούτε πολιτική βούληση, ούτε κότσια, ούτε πολιτικό θάρρος. Ευτυχώς που υπάρχει και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Ιντβέλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πρέπει να είμαι ιδιαίτερα σύντομη και ζητώ συγγνώμη, θα πρέπει να φύγω αμέσω μετά. Αλλά δέχομαι όσα είπε ο Μάικλ κατά λέξη είναι απαράδεκτο, απαράδεκτη η μεταχείριση ορισμένων κρατών μελών και η δικαιολογία που προβάλλουν, γιατί όταν μιλάνε για ίση μεταχ... ότι η ίση μεταχείριση ανθρώπων με αναπηρία ίσως είναι κάτι το ιδιαίτερο δαπανηρό, μα δείτε τι δαπανούμε για ανοησίες. Αν δω τη δική μου έκθεση για την καταπολέμηση τρομοκρατίας, το κόστος αυτό έχει αυξηθεί κατά 20 φορές τα τελευταία 10 χρόνια και μερικοί δεν θέλουν καν να δουν τις δαπάνες, διότι λένε είναι ότι τόσο σημαντικό θέμα που δεν έχει σημασία πόσα δαπανούμε. Γιατί τότε μιλάμε για καταπολέμηση της τρομοκρατίας και όχι την προστασία των πολιτών της Ευρώπης. Κύριε Μποσκούρτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Παρακολουθώ το θέμα αυτό ήδη από το 2008 εξ Σοσιαλιστών και Δημοκρατών αλλά διερωτώ με μετά από αυτά που ακούσαμε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, τι γίνεται. Υπάρχει προθυμία να ασχοληθούμε με τις διακρίσεις. Κοιτάω το σχέδιο που αναφέρεται σήμερα. Μόνο για τους ε, ανθρώπους με αναπηρία ε, μιλούν. Αλλά ε, πρόκειται και για άλλους, και άλλες διακρίσεις και με βάση την ηλικία, το γενετήσιο προσανατολισμό ή τη θρησκεία τι κάνουμε. Όποτε το συζητούσαμε στο κοινοβούλιο όλοι λέγανε ότι είναι α, πολύ ακριβό, πολύ ακριβό, ειδικά για την αναπηρία. Τώρα ασχολούνται με την αναπηρία. Μπράβο, λαμπρά και θαυμάσια. Για τους υπόλοιπους λόγου, τι γίνεται. Ή δεν η πρόφαση επειδή ασχοληθήκαμε με την αναπηρία τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη. Υπάρχει προεθυμία λοιπόν να το κοιτάξουμε το θέμα αυτό. Και το δεύτερο, στη συζήτηση που έγινε με την Επίτροπο, κυρία Ρέντινγκ, πριν από κάποιο διάστημα, είπε ότι, α, κοιτάξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα, εντάξει, και οι άλλες αιτίε, μήπως πρέπει να κάνουμε μια οδηγία ξεχωριστή για την αναπηρία. Αυτά που λέει σήμερα το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών, τα έχουμε αφήσει στην άκρη όλα τα άλλα. Ο κύριος Ντουγιόγκ, στα αγγλικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Απολύτως. Είναι έσχος. Και επίσης ε, κρίμα που η Προεδρία αναφέρθηκε μόνο σε ένα λόγο διακρίσεων και δεν ε, ασχολήθηκε με τους υπολείπους. Στο Κοινοβούλιο είναι σαφές ότι θέλουμε την οδηγία αυτή και ε, δεν καταλαβαίνουμε καθόλου γιατί πρέπει να περιμένουμε τόσο πολύ καιρό για να γίνει οποιαδήποτε πρόοδος. εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική βούληση και τίποτα άλλο. Επίσης, θα μιλήσει ο κόσμος και συγκεκριμένα ο δρόμος. Έχω ξεκινήσει στην Ολλανδία μια δράση με τη βοήθεια ε, των οργανώσεων ομοφιλοφίλων, ε, λεσβιών ε, και λοιπά και για τα δικαιώματά τους. Active λέγεται οργάνωση και μια εφημερίδα που έχουν και ζητούμε από όλους κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών να σημειώνουν οποιοδήποτε είδος διάκρισης και μη διαπιστώνουν ε, είτε εναντίον τους είτε εις βάρος άλλων ε, γνωστών τους που θα συναντήσουν στις διακοπές και ελπίζω να υπάρξει μεγάλος φάκελος αποδείξεων για να δείξουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη και πραγματική ανάγκη. Και ενδεχομένω και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι από το Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο στη χώρα τους και να συνενώσουμε όλες τις αποδείξεις το τι συμβαίνει στην καθημερινή πράξη για να καταλάβει η επόμενη Προεδρία ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοια έσχη με την παρούσα. Ευχαριστώ. κυρία Ačiū labai. Iš tikrųjų labai blogai, kad e, taip lietai judam į priekį dėl labai... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ κρίμα πραγματικά το γεγονός ότι γίνονται τόσο αργά βήματα σε μια τόσο σημαντική οδηγία για τους πολίτες. Ε, μια προεδρία αντιγράφει την άλλη. Ή μάλλον υποδίεται ότι εργάζεται, ότι το ψάχνει, ε, επιλέγει ένα λόγο διακρίσεων εργάζεται σε αυτό το φάκελο ή υποκρίνεται ότι εργάζεται, ε, αλλά μηδέν στο πηλίκον. Είναι σημαντικό και τα άτομα με αναπηρία να έχουν παντού τα ίδια δικαιώματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ωραία. Υπάρχει όμως μια έκθεση για την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία. Και χαίρομαι που είναι παρόν και ο εισηγητής. Και τρεις πολιτικές ομάδες, οι πράσινοι, οι σοσιαλδημοκράτες και άλλη μία που είναι η φιλελεύθερη, είναι υπέρ ε, της ταχείας έγκρισης ε, της οδηγίας αυτής. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ακόμα να μας υποστηρίξει. Καταλαβαίνετε πόση σημασία δίνει το ΕΛΚ στους ανθρώπους με αναπηρίες. Ε, όλοι θέλουμε να ληφθεί μια απόφαση επιτέλους. Και εμείς οι πολιτικοί να μην εμφανιζόμαστε μόνο ε, στις προεκλογικές εξαρτίες και να είμαστε σε επαφή με αναπήρους. Κύριε Βέξτραμ, και εγώ είμαι εξίσου εκνευρισμένη και εξοργισμένη με τους προλαλήσαντες, τον κύριο Κάσμαν και άλλους ελάχιστα γίνονται σε σχέση με αυτό το σημαντικό θέμα. Σε ό,τι αφορά τις αναπηρίες, υπάρχει η σύμβαση του ΟΗΕ που έχει τεθεί σε ισχύ από φέτο τον Ιανουάριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξασφαλίζει τα δικαιώματα σε ανεξάρτητη διαβίωση και αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους και τον τρόπο διαβίωση και η πρόσβαση σε στοιχειώδεις ε, υπηρεσίες πρόνοιας είναι σημαντικό ζήτημα που αναφέρεται σε αυτή τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ανθρώπων με αναπηρίες. Και πώς χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά κονδύλια για υπέρ των αναπήρων. Οι κυβερνητικέ οργανώσεις μας έχουν επισημάνει ότι εκείνες ε, χρηματοδοτούν ε, τα κτίρια ε, Προσφορά τέτοια κοινωνική πρόνοιας που τελικά καταλήγουν σε περιθωριοποίηση και όχι στην αναμενόμενη ένταξη. Είναι μια πραγματικά κακή χρήση των ε, διαρθρωτικών κονδυλίων που θα πρέπει να χρηματοδοτούν την πρόθεση ανεξάρτητης διαβίωσης των αναπήρων και όχι την ε, εισαγωγή τους σε ιδρύματα. Επίσης το θέμα της ανθρώπινης μεταχείρισης των αναπήρων στα, στους διάφορους, στα διάφορα ιδρύματα και Επαναλαμβάνω την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ανεξάρτητη διαβίωση των αναπήρων, στη διεκδίκηση της ανεξαρτησίας τους και θα ήθελα να ενθαρρύνω το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της χρήσης αυτών των διαρθρωτικών κονδυλίων. Κύριε Ρωμέβα, είστε εισηγητής. Ακούσατε τα σαφή και πολυτολμηρά σχόλια των μελών της Επιτροπής μας και έχετε το χρόνο για λίγα σύντομα τελικά σχόλια πριν υποδεχθούμε την κυρία Λεμπάγη. Δύο λόγια μόνο, ήταν σαφέστατο το μήνυμα. Όλοι όσοι έλαβαν το λόγο μίλησαν ε, για αυτό το θέμα και νομίζω ότι να έλαβε, να, ελπίζω να έλαβε το μήνυμα και η Επιτροπή και η Προεδρία και το Συμβούλιο. Περιμένουμε ακόμη αυτή την έκθεση το συντομότερο δυνατό και για το περιεχόμενο αλλά και για την νομική υποχρέωση που φέρουμε για την ε, έκθεση αυτή. Δεν το αντελήφθη φαίνεται αυτό η Ουγγρική Προεδρία. Ελπίζω η Πολωνική Προεδρία να το καταλάβει, να το κατανοήσει καλύτερα. Και ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που έχουμε τόσο τέτοιες ε, συζητήσεις με εκνευρισμό και οργή. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα κληθούμε να συζητήσουμε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε κιόλα. Ευχαριστούμε. Τώρα θα γίνει μια ενημέρωση από την κυρία Λεμπάγι για τις συμφωνίες ότι αφορά την προστασία δεδομένων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ενημέρωση αυτή από την κυρία Λεμπάη θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, οπότε παρακαλώ όσοι δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε κεκλεισμένα των θυρών συνεδριάσεις, παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα και εμείς να υποδεχθούμε την κυρία Λεμπάγ. Καλώς ήρθατε κυρία Λεμπάγ. Έχουμε ξεπεράσει και το ωράριο της διερμηνίας. Οπότε απελευθερώνω και τους διερμηνείς. Μπορούμε την κεκλεισμένα το θερό συνεδρίαση να την κάνουμε και χωρίς διερμηνία. Καλό σας μεσημέρι.